Dear colleagues, good morning. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ας αρχίσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Με ιδιαίτερη χαρά Καλωσορίζω εδώ την κυρία Βιέρα Γιούροβα, η οποία είναι η υπεύθυνη για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων, για να ανταλλάξουμε απόψει στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου της Επιτρόπου με την Επιτροπή μας. Κυρία Γιούροβα, έχουμε θέματα που εκρεμούν ακόμα και πρέπει να ολοκληρωθούν, όχι όμως μόνο αυτό, Ελπίζουμε εσείς να έχετε όσο γίνεται περισσότερα αποτελέσματα πριν από τη λήξη της αυτής. Σας δίνω λοιπόν ε, το λόγο, χωρίς άλλη καθυστέρηση, για να μας παρουσιάσετε τα θέματα που έχουμε ακόμα μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, λέει η κυρία Γιούροβα. Όντως, ε, ακόμα έχω αποτελέσματα να προσφέρω. Αύριο θα εγκρίνουμε μεγάλο πακέτο για τις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο εδώ και καιρό. Οπότε από τη δική μας την πλευρά αυτό θα κάνουμε. Χτες ήταν οι καταγγέλλοντες, οι συλλογικές ε, αποζημιώσεις, θέματα για τους καταναλωτές πολύ σημαντικά. Όντως, έχουμε κοινό έργο. Η Επιτροπή σας και εμείς και γι' αυτό πολύ χαίρομαι που μπορούμε να έχουμε αυτό το διάλογο μεταξύ μας. Όπως σας είπα, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα, τώρα που έχουμε εγκρίνει την αυτή συμφωνία για τους καταναλωτές. Νέα πρόταση που έχει να κάνει με τις λογικές αποζημιώσεις και το αστικό δίκαιο στην Ευρώπη. Και αυτό, αφότου έχουμε εγκρίνει και την πρόταση για τους καταγγέλλοντες, κάτι το οποίο σας παρουσίασε χτες ο κύριος Τίμερμανς που ήταν εδώ. Και πριν ε, εγκρίναμε και ένα μεγάλο πακέτο για τις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο ήθελε και η Επιτροπή σας. Τώρα, πολύ σύντομα θα πω στις λεπτομέρειες. Πρώτα απ' όλα, η νέα πρόταση για τις λογικές αποζημιώσεις. Εργαζόμαστε από το 2013 με τη σύσταση που υπήρχε για το θέμα αυτό, κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές στην Ευρώπη όταν πρόκειται για τα δικαιώματα των καταναλωτών και πώς αυτά προστατεύονται. Τώρα όμως φάνηκε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσουμε. Και έτσι βασιστήκαμε στη σύσταση του 2013 για τις λογικές αποζημιώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσουμε στο μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι. Δεν πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις δικηγόρων κτλ. Εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε κάποιες ρήτρες ασφάλειας κατά των καταχρήσεων. Εμείς θέλουμε πλήρη διαφάνεια και έλεγχο της χρηματοδότησης από τρίτα μέρη. Έχουμε αφήσει πριό στις χώρες ε, μέλη, ώστε να μπορούν ε, επίσης να δράσουν βάσει των δικών του συστημάτων αστικού δικαίου. Οπότε βασίζομαι στη δικιά σας στήριξη για να συνεχίσουμε να εστιάζουμε σε αυτήν τη σημαντική πρόταση, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις πριν από τις επόμενες εκλογές. Οι υπηρεσίε μου και εγώ να ξέρετε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε και να ξέρετε ότι και το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα ως προτεραιότητα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Χθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και πρόταση για οδηγία προκειμένου να ενισχύσει την προστασία των καταγγελόντων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε το LuxLeaks, Panama Leaks ε, ή το Cambridge Analytica τελευταία. Όλες αυτές οι περιπτώσεις κατέδειξαν πόσο σημαντική είναι η παρουσία των καταγγελόντων στην σημερινή σύγχρονη οικονομία μας. Και είμαι ευγνώμων για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό το θέμα, κυρίως ε, συγκεκριά σας. Χτες ακούσατε τον ε, Αντιπρόεδρο για την πρόταση αυτή. Θέλαμε να παρουσιάσουμε ε, υψηλή ποιότητα, κοινέ προδιαγραφές για την προστασία των καταγγελόντων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Επίση, φροντίσαμε να υπάρχουν οι κατάλληλοι δίωδοι, ώστε οι καταγγελίε αυτές να μπορούν να γίνουν πρώτα απ' όλα σε εσωτερικό επίπεδο, με εσωτερικέ διόδου, μετά με εξωτερικέ διόδου και μετά απέναντι στο κοινό, στους δημοσιογράφους. Πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες εκθέσεις, να υπάρχει feedback στους καταγγέλλοντες. Τα αντίπεινα απαγορεύονται κατά των καταγγελόντων. Αντίθετα, πρέπει να υπάρχουν συστήματα προστασίας τους. Η πρότασή μας έχει ως στόχο να προστατεύσει την υπεύθυνη καταγγελία, ακριβώς για να προστατευτεί το κοινό καλό. Συγχρόνως η οδηγία συμπεριλαμβάνει ρήτρες ασφάλειας για να αποθαρρύνονται οι περιπτώσεις ε, καταγγελιών που γίνονται εκ του πονηρού. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια ισορροπημένη προσέγγιση. Αύριο η Επιτροπή θα κάνει ένα ακόμα βήμα για μια ε, δίκαιη εσωτερική αγορά μετά από όσα έχετε εσείς ζητήσει αλλά και οι χώρες μέλη. Ανταποκρίνεται όμως και στη ζήτηση που υπάρχει από τις επιχειρήσεις, από τους εταίρους μας για νομική βεβαιότητα. Κυρίως μετά την απόφαση την πρόσφατη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την υπόθεση Πόλμπουτ. Εμείς έχουμε ευαισθητοποιηθεί και υπό το φως όλων αυτών Τώρα προτείνουμε σύγχρονου και δίκαιου κανόνε για την κινητικότητα των επιχειρήσεων μέσα στην εσωτερική αγορά. Και για πρώτη φορά προτείνουμε κανόνε για την διασυνοριακή κατανομή. Θέλουμε οι τίμοι επιχειρηματίε να μπορούν πλήρω να αποφεληθούν από την εσωτερική αγορά. Γι' αυτό και έχουμε συμπεριλάβει ρήτρε ασφάλεια για τι μειονότητε, για του πιστωτέ κτλ δεν θέλουμε τεχνητούς ε, διακανονισμούς, ούτε επιχειρήσεις που είναι μόνο μία θηρίδα. Θέλουμε να εξυγχρονιστούν οι επιχειρηματικοί κανόνες. Η πρόταση για τα ψηφιακά θα προσφέρει στις επιχειρήσεις λύσεις για αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Θα βοηθήσει τις σχέσεις μεταξύ τους και με χαμηλότερο κόστος προβλέπονται και ρήτρες ασφάλειας κατά των καταχρήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ακαιρεότητα και η αξιοπιστία των διαδικασιών online. Τα ψηφιακά μέσα θα προσφέρουν και περισσότερη διαφάνεια. Επ' αυτού λοιπόν βασίζομαι στη δική σας στήριξη. Ελπίζω ότι το έργο για την πρόταση αυτή θα αρχίσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για την νομοθετική αυτή πρόταση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές και σκιώδες συνεισηγητές για την δικιά του συνεισφορά ε, όσον, αφορά την πρόταση για τις ψηφιακές συμβάσεις. Συναντήθηκα με όλους τους συνεισηγητές την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Και πραγματικά με ενθαρρύνουν οι πραγματικές προσπάθειες των κ. Φως και Γκέπχαρτ προκειμένου να καταλήξουμε σε πρακτικές λύσεις είναι ευέλικτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι διατεθειμένη να βοηθήσει τους συνομοθέτες να καταλήξουν σε συμβιβασμούς επί των προτάσεων αυτών. Η κοινή μας ε, στόχη πρέπει να είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την πρόταση όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας και να προχωρήσουμε και όσον αφορά την πώληση αγαθών ε, στα πλαίσια της επόμενης Προεδρίας και έτσι να έχουμε συμφωνία και από αυτού. Μια άλλη υπόθεση τώρα όπου μπορούμε να προχωρήσουμε είναι εκείνη για την αφεγγερότητα. Να ξέρετε πάντως ότι οι υπηρεσίες μου θέλουν να βοηθήσουν την Επιτροπή σας προκειμένου να υπάρξει απόφαση σε πρώτη ανάγνωση πριν την, τις επόμενες ευρωεκλογές. Πρέπει να υπάρξει μεγάλη φιλοδοξία όσον αφορά την πρόταση αυτή, κυρίως για να βοηθήσουμε και τους επιχειρηματίες, αλλά κατά πρώτον αυτούς που χρωστάνε. Να ξέρετε ότι θα γκρίνουμε επίσης πρόταση για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως πολύ σωστά αναγνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες για να επηρεάσει πολλές πτυχές στις ζωές μας. Και είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθεί η τεχνητή νοημοσύνη με το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για να προωθήσει την καινοτομία αλλά συγχρόνως να σέβεται τις αξίες της ε, Ένωσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Επιτροπή λοιπόν θα προτείνει μια συνολική προσέγγιση για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η ερευνητική αριστεία. Να θέσουμε τις βάσεις για ένα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο και να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των πολιτών για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία έχει προχωρήσει όσον αφορά την ηθική για την ε, τεχνητή νοημοσύνη και πιστεύουμε ότι θα καταλήξουν στα τέλη της χρονιάς αυτής. Ανοίγουμε την πόρτα επίσης για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα περί ευθύνης. Το 2019 η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τις ευρύτερες επιπτώσεις ε, των κενών και του προσανατολισμού όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, το ίντερνετ ε, των πραγμάτων και την ρομποτική. Τα πρώτα αποτελέσματα όμως για την τεχνητή νοημοσύνη ελπίζουμε ότι θα θέσουν τη βάση για τον ε, σωστό ανταγωνισμό και να μπορέσουμε έτσι να είμαστε σε ηγετική θέση στην παγκόσμια σκηνή. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, είμαι πεπισμένη ότι συνεχίζοντα τη στενή συνεργασία μεταξύ μα, οι προσπάθειές μα θα καρποφορήσουν και θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα στην επόμενη χρονιά. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και Προσβλέπω στις δικές σας απόψεις και ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Επιτροπέ, για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και έχω τέσσερις ε, συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Χάουτα, πρώτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, Επιτροπέ. Καταρχάς, ε, για αυτά τα θέματα για τις ε, πωλήσει τις επιγραμμικές από των αγαθών. Ξέρετε ότι ήταν πολύ απογοητευτικό το αποτέλεσμα της Επιτροπής μας σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν ε, υπήρξε πλειοψηφία ούτε για την ε, ελάχιστη ούτε τη μέγιστη αρμόνιση της προστασίας του καταναλωτή. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι μπορεί να επιληθεί η κατάσταση προκειμένου κανένα κράτος μέλος να μην διακυβεύσει την ίδια επιτευχθήσα ε, προστασία του καταναλωτή. Ενδεχομένως να υπάρξει μια κατάσταση ε, κατοχύρωσης των επιτευγμάτων χωρίς δυνατότητα ε, βελτίωσης. Αυτό θα με ανησυχούσε όμως ιδιαίτερος, γιατί θα ήταν πάρα πολύ άδικο για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που μπορεί να μην έχουν αναβαθμίσει ακόμα την προστασία καταναλωτή. Δεύτερη ερώτηση, γιατί είδα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα σχέδιο δράση για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Γιατί είναι χρηματοδοτική αρρωγή σε ό,τι αφορά την ατζέντα για το κλίμα και για την βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στο σχέδιο δράση ότι θα υπάρξει fitness check για την νομοθεσία και τη ε, υποβολή αναφορών σε ό,τι αφορά και την οδηγία για τη δημόσια χρηματοδότηση και έγινε και μια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς για να εκτιμηθεί η ανάγκη τα συμβούλια των εταιριών να έχουν πρόσβαση σε σωστή α, χρηματοδότηση και να υπάρχει και σωστή και ιδέουσα επιμέλεια στα θέματα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι η υπηρεσία σα και εσεί προσωπικά παίζετε σημαντικό ρόλο για να εφαρμόσουν όλα αυτά που θα αποτελέσουν και τμήμα α, των οδηγιών του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή και σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και τέλο να σα πω ότι η πρόταση για τι συλλογικέ αγωγέ που παρουσιάσατε προσφάτω θα μπορούσε και αυτή να παίξει ρόλο για την εφαρμογή των δικαιωμάτων, ε, μάλλον την ε, πραγματοποίηση και την υλοποίηση των δικαιωμάτων των θυμάτων ε, μεγάλων εταιριών σε ό,τι αφορά και ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς συμβάσεις και επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής θεωρώ ότι θα βελτιώσουμε τα δικαιώματα των θυμάτων. Δυστυχώ η πρόταση περιορίζεται στα δικαιώματα των θυμάτων των καταναλωτών. Γιατί έγινε αυτή η επιλογή θα ήθελα να ρωτήσω. Ε, Κυρία Ραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε και καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρόταση για τους πληροφοριοδότες. Αυτό αποτελούσε επικαιρό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πραγματικά εδώ επιδείξατε ηγετικέ ικανότητα και κάνατε μία πρόταση η οποία καλύπτει πολλού τομεί τη ευρωπαϊκή πολιτική. Θα ήθελα να μα πείτε πώ του επιλέξατε αυτού του τομεί. Γιατί είναι ευρεία η πρόταση, αλλά δεν είναι αρκετά συνεκτική. Υπάρχουν τομεί τη Ευρωπαϊκή αρμοδιότητα όπου η οδηγία δεν θα ίσχυε. Αυτό προκαλεί μια έκπληξη και μεγάλη σύγχυση και για του πληροφοριοδότες. Ένα παράδειγμα να σα δώσω, στην ενέργεια για παράδειγμα η ασφάλεια των πυρηνικών εργοστασίων θα καλύπτονταν από την οδηγία, αλλά όχι η ασφάλεια των ε, εργοστασίων άνθρακα. Είναι δύσκολο από πλευρά ε, πληροφοριοδοτών να ξέρουν κατά πόσο καλύπτονται ή δεν καλύπτονται από την πρόταση αυτή. Καταλαβαίνω ότι μια εντελώς οριζόντια πρόταση που θα καλέψει και τα, μέλη, τα αποτελεί πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον θα περίμενα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιλάμβανε όλους τους τομείς που μπορεί να περιλάβει για να καταλήξουμε σε μια πρόταση η οποία θα είναι όσο το δυνατόν πιο εγκάρσια γίνεται. Να συμφωνήσω και με αυτά που είπε η κυρία Χάουταλα για τις συλλογικέ αγωγές. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα και για τις δύο προτάσεις, γιατί, ξέρετε, κατά κάποιο τρόπο αλληλοσυμπληρώνονται συμπληρώνονται. Η πρόταση για τους πληροφοριοδότες ελπίζουμε ότι θα αποκαλύψει πιο πολλά θέματα που απασχολούν τους καταναλωτές και στη συνέχεια να ακολουθήσει η συλλογική αγωγή όπου αυτό είναι απαραίτητο. Και νομίζω λοιπόν ότι και οι δύο προτάσεις θα πρέπει να είναι το δυνατόν ευρύτερε. Μία ερώτηση έχω να κάνω για την πρόταση για το ψηφιακό περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε. για το Κοινοβούλιο και την προθυμία που επιδεικνύει να ολοκληρωθεί αυτή η πρόταση των Συντομετρών δυνατών. Αλλά ένα από τα πιο βασικά προβλήματα είναι το θέμα του διαδικτύου για τα πράγματα, για το Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ απαραίτητο αυτό, γιατί αν εξαιρεθεί το Internet of Things, το διαδικτύο των αντικειμένων, δεν μας καλύπτει δεν μας καλύπτει και η απάντηση ότι θα καλυφθεί από μετέπειτα πρόταση το διαδίκτυο των αντικειμένων α, για την πώληση δηλαδή των αγαθών. Γιατί στο διαδίκτυο των αντικειμένων η πώληση αντικειμένων πλέον αποτελεί όλο και πιο μικρό μερίδιο. Πιο πολύ περνάμε σε leasing, σε ενοικίαση και διάφορες μορφές μίσθωση για αυτοκίνητα ή για παράδειγμα ε, σύμβαση άμα παραχής υπηρεσιών για το ψυγείο του καθενός και όταν τελειώσει η σύμβαση επιστρέφεται το αντικείμενο. Αν δεν καλυφθεί λοιπόν το διαδίκτυο των αντικειμένων στην πρόταση αυτή, θα μείνει ένα πλάτος τελείως ακάλυπτος, γιατί η πρόταση για την πώληση αγαθών δεν θα καλύψει αυτό το μεγάλο κομμάτι. Άρα, θέλουμε να υπάρξει πραγματικά κίνηση από πλευρά ε, Επιτροπής, της Επιτροπής και του, και του Συμβουλίου για να καλυφθεί το διαδικτύο των αντικειμένων. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να ξεπεράσετε αυτό το μεγάλο εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας για την ψηφιακή πρόταση. Ευχαριστώ κυρία Ρίγνερ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, είναι πραγματικά συναρπαστικό να σας ακούμε προς το τέλος της θετίας ε, γιατί τότε είναι που ξεπηδούν τα πραγματικά συναρπαστικά αντικείμενα. Και φυσικά οι πληροφοριοδότες είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε πολύ και για το οποίο πολεμήσαμε και για τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Ε, όλα αυτά λοιπόν είναι συναρπαστικά θέματα και πιστεύουμε και ελπίζουμε μάλλον να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε και μέχρι το τέλος της θητείας. Μία ερώτηση. Πώς φαντάζεστε το χρονοδιάγραμμα εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως βουλευτές. Ε, θα κάνουμε φυσικά ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιληθούν τα ζητήματα αυτά, αλλά το Συμβούλιο γενικά είναι πολύ πιο αργό. Πρόκειται να βιαστεί. Και επίσης ε, θα καταφέρουμε να τελειώσουμε αυτά μέχρι το τέλος της θητείας. Για το πακέτο για το εταιρικό δίκαιο. Έχουν ρωτήσει κάτι. Και εδώ η Επιτροπή θα πρέπει να κοιτάξει να κάνει μια πρόταση για την κινητικότητα των εταιριών, η οποία είναι απαραίτητη. Αλλά προφανώ χρειάζεται θάρρο, γιατί όταν πρόκειται για θέματα αστικού δικαίου και εργασιακά, όλοι ξέρουμε πόσο καιρό παίρνουν τα πράγματα και ότι πολλά ζητήματα ε, επιφέρουν μεγάλες ανασφάλειες, οι οποίες πάντα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Άρα, το πακέτο, τι ασφάλεια προσφέρει για το forum shopping για να αποδειχθεί η μεγαλύτερη κινητικότητα των εταιρείων. Και έχω υπόψη μου για κάποιες ελάχιστες προτεγραφές κάποιες προτεγραφές ε, για ελάχιστο κεφάλαιο, αποφυγή των, των πρακτικών ε, φοροαποφυγής. Τα ξέρετε όλα αυτά. Και προφανώς θα πρέπει να ασχοληθούμε και με όλα αυτά τα θέματα, προκειμένου το πακέτο αυτό, το οποίο προφανώς ε, και το καλώς ορίζουμε, αλλά όλες αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες θα πρέπει να είναι στη θέση τους ε, πρωτού ξεκινήσουμε την νομοθετική εργασία. Μία άλλη ερώτηση. Αυτές οι προτάσεις σε τι βαθμό συνάδουν με τις ιδέες του κυρίου Γιούνκερ για μια πιο κοινωνική Ευρώπη είναι συμπατές. Μήπως δεν χρειάζεται ένα αντιστάθμισμα αυτή η κινητικότητα των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά δηλαδή το δικαίωμα στην απόφαση των εργαζομένων για να υπάρχει αντιστάθμιση του δικαιώματος και φυσικά το πακέτο για, την, ε, για το δίκαιο των εταιριών πώς θα δημοφορτεί μέχρι το τέλος της Ευχαριστώ κύριε Σουσάμι uh, uh, to... Ευχαριστώ. Συμφωνώ, Επίτροπε, με τους συναδέλφους. Ε, εκτιμώ το γεγονός ότι ακούσατε τις διάφορες εκκλήσεις που έχουμε κάνει για διάφορα θέματα και κυρίως για το θέμα των καταγγελόντων. Η ανακοίνωση της Επιτροπής χθε ότι πήρε απόφαση να ενισχύσει τα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτη. Και τώρα θα πρέπει να συνεχίσουμε αμελητή επ' αυτού θέματος. Θέλω να συνδέσω το ρόλο των πληροφοριοδοτών με την μαλτέζικη εμπειρία για τους ρεπόρτερ. Γιατί και μέσω της δράσης αυτών ε, γνωρίζει διάφορα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα το κοινό. Στο έγγραφο της Κομισιόν, το Fact Finding Sheet, μιλάτε για την προστασία των καταγγελόντων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μαλτέζικη εμπειρία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι το ιδιάζον. Γιατί εάν ένας πληροφοριοδότης στη χώρα μιλήσει για ένα θέμα το οποίο αρέσει στην ε, κυβέρνηση, τότε προστατεύεται. Και του δίνουν και διάφορες συμβόλαια και συμβάσεις. Εάν όμως ήταν, είναι ένα άτομο, όπως η Φίμωβα, ε, η οποία έκανε κάποιες δηλώσεις για την τράπεζα Πιλάτους, για θέματα ξεπλήματος χρήματος, αυτό το άτομο δεν προστατεύεται και μάλιστα κινδυνεύει. Ε, υπήρχε και θέμα εκδοσής της μάλιστα. Και αυτό ε, συνδέεται με αυτό που είπατε στην αρχή, για τον εντοπισμό των αρχών που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις περιπτώσεις των καταγγελόντων. Αυτές οι αρχές, εκτός από το ότι αντιμετωπίζουν την υποχρέωση ε, υποβολής εκθέσεων, πρέπει να είναι και ανεξάρτητες. Γιατί οι αρχές οι οποίες δίνουν ε, το καθεστώς ας πούμε, του καταγγέλλοντα, μερικές φορές έχουν συμφέρον να το δώσουν, να μην το δώσουν. Και επομένως, ε, νομίζω ότι εκεί θα καταρρεύσει το σύστημα. Ε, και επίσης διάβασα από το, την εφημερίδα Times of Malta ότι θα είσαστε στη Μάλτα τον Ιούνιο. Ε, θα έρθετε στη Μάλτα τον Ιούνιο. Ε, και η ώρα η Κομισιόν να προστατεύσει τα συμφέροντα των ανθρώπων και να το δει αυτό ο κόσμο στη Μάλτα. Ε, φαντάζομαι θα εξετάσετε και διάφορα θέματα τα οποία αφορούν άτομα, τα οποία είναι υπεύθυνα. Για το θάνατο της ε, δημοσιογράφου της Μαλτέζας δεν έχουν ε, διωχθεί ακόμα. Όλα τα μέτρα λαμβάνονται, το συντομότερο δυνατό φαντάζομαι, όχι μόνο για την καλύτερη προστασία των καταγγελόντων, αλλά και για θέματα ξεπλήματος χρήματος και την, θέματα συναφή με την οδηγία για το ξεπλήμα του χρήματος. Φαντάζομαι ότι θα το συζητήσουμε και αυτό στη Μάλτα. Γιατί αν κοιτάξετε την εξέλιξη της οδηγίας, βλέπετε και τη σημασία που έχει αυτό το θέμα ε, για τις αποκαλύψεις, ειδικά του, για την τράπεζα Πιλάτους. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Να σας συγχαρώ και εγώ, όπως και οι συνάδελφοι. Δυστυχώς όμως ξέρετε ότι κάποια μέλη του Κοινοβουλίου περιμένουν ανυπόμονα την ανακοίνωση για την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, το πρώτο μου ερώτημα θα ήταν να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Γιατί πισέρχονται διάφορες γενικές διευθύνσεις εδώ που είναι συνυπεύθυνες. Καλώς ορίζω και αυτόν τον οδηγό που μας, ή τον οποίο μας μιλήσατε, που θα είναι έτοιμος μέχρι το τέλος του χρόνου. Το άλλο θέμα είναι το θέμα της ευθύνης. Εκεί μιλήσατε πολύ διστακτικά και προσεκτικά. Είπατε ότι ανοίγετε την πόρτα για μια λύση. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα λύση για το θέμα της ευθύνη. Το ερώτημά μου είναι, δεν φοβάστε ότι τα κράτη-μέλη θα υποβάλουν σχετική εθνική νομοθεσία. Κάποια κράτη-μέλη είναι πολύ δραστήρια σε αυτό το τομέα και προωθούν κανόνες δικούς τους. και αυτό δυσκολεύει το έργο των Ευρωπαίων συνομοθετών. Τι θα κάνετε ούτως ώστε να ασχοληθείτε εσείς με αυτό το θέμα για να εμποδίσετε ένα κατακαιρματισμό του, του κανονιστικού πλαισίου. Ενημερώθηκα μάλιστα ότι και σε επίπεδο ΩΣΑ υπάρχουν ανησυχίες ότι και για τα, τις δοκιμές και τα πιλωτικά προγράμματα για τα αυτόνομα οχήματα, οι διαφορετικές χώρες, διάφορες δικαιοδοσίες έχουν διαφορετικές ε, προσεγγίσεις. Ακόμα και για τις δοκιμές είναι δύσκολο να έχουμε ενιαία προσέγγιση. Διερωτώμε πώς θα έχουμε ενιαίο και κατάλληλο πλαίσιο για όλα τα θέματα των αυτόνομων οχημάτων, εάν κολλάμε ήδη στις δοκιμές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα ε, για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία δεν θέλει κατακαιρματισμένη αγορά. Ευχαριστώ κύριο Καβαντά, ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ένα γρήγορο σχόλιο και ένα ερώτημα. Το σχόλιο είναι ότι είμαι πολύ ικανοποιημένο κι εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, που ασχοληθήκατε με το θέμα των καταγγελόντων που δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητο μέσα σε αυτό το χάος σκανδάλων που ξεσπούν το ένα μετά το άλλο. Θέλω να εστιάσω σε δύο σημεία από αυτού. Με μεγάλη προσοχή θα, θα ασχοληθώ με το θέμα της προστασίας των πηγών και των δημοσιογράφων από την άλλη. Όταν πρόκειται για ευαίσθητα θέματα, όπως είπε προηγουμένως και ο Μαλτέζος συνάδελφος. Παρενθετικά, εκπλήσουμε που δεν έχουμε πραγματικό εργαλείο για να καταγγείλουμε το μαλτέζικο κράτος, που ξέρουμε ότι υπάρχει διαφθορά στο υψηλότερο επίπεδο. Ε, μιλάμε δηλαδή για, την, για μια συμπεγνία ανάμεσα σε υπουργού και στους εντολοδότες της δολοφονίας. Εμείς τι κάναμε, ένα ανακοινοθέν, μια διαμαρτυρία. Είναι ανεπαρκές. Θα πρέπει να δούμε τις επόμενες φάσεις τώρα γιατί προς το κοινό συμφέρον θα πρέπει να τιμωρήσουμε ένα κράτος ένοχο, συνένοχο για μία δολοφονία. Υπάρχουν αποδείξεις, παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία δικαστική απόφαση. Ένα μέλος της κυβέρνησης, τουλάχιστον της Μάλτας, εμπλέκεται. Το κείμενο που παρουσιάσατε Κυρία Επίτροπε, ε, για τους καταγγέλλοντες, το παρουσίασε ενδελεχώς χθε ο κύριος Τίμερμαντς, ε, τον οποίο δεν άκουσα γιατί υπήρχε πρόβλημα με το τρένο μου. Αλλά ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε στα άκρα, να ανοίξει το κουτί τη πανθόρας και να μπορούμε να το κλείσουμε. Το βασικό είναι να εξασφαλίσουμε πραγματική ε, προστασία για του ανθρώπου που κάνουν πράγματα για το κοινό καλό. Και το κείμενο αυτό είναι ένα καλό συμβασμό ανάμεσα στα δύο άκρα. Ε, είναι μια καλή δουλειά, είμαι ικανοποιημένο όπω και άλλοι συνάδελφοι. Ένα άλλο τώρα θέμα, μια ερώτηση, είναι πολύ απλή ερώτηση. Έφερε αντιμέτωπο αυτό το θέμα απέναντι στον κύριο το Κοινοβούλιο απέναντι στον κύριο Εμίλιο Κατάνη για μία απόφαση. Για μία υπόθεση ΤΕΣ 140 κάθετος 15, για μία διαβόητη υπόθεση που αφορά τη δημοσίευση των τετράστιλων κειμένων που χρησιμοποιούμε στους τριλόγους. Καλή είναι η διαφάνεια, αλλά αν γίνει ακραία, σε τέτοιο βαθμό που σε όλες τις φάσεις ένα κείμενο θα πρέπει να δημοσιοποιείται, τότε πρέπει να σκεφτούμε το νέο ρόλο που θα προσφέρουμε στα λόμπι. Θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν μέρος στις διαπραγματεύσεις και μπορούν να τι παραλύσουν τις διαπραγματεύσεις. Θα δεχτείτε την απόφαση αυτού, αυτή του δικαστηρίου, θα κάνετε προσφυγή εναντίον αυτής της απόφασης, όπου προσέφυγε δηλαδή το Κοινοβούλιο εναντίον του κ. Κατάνη, μάλλον ο κ. Κατάνη εναντίον του Κοινοβουλίου. Ο επόμενο ομιλητή. Θέλω να συγχαρώ και εγώ την Επίτροπο, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Παρουσιάσατε το πακέτο που συζητάμε σήμερα. Αν το είχατε παρουσιάσει στην αρχή της θητείας μας, θα ήταν πολύ καλύτερο. Κάνατε μια τεράστια δουλειά βέβαια και δυστυχώς έρχεται αυτή τη χρονική στιγμή, τη στιγμή δηλαδή που έχουμε μόνο ένα χρόνο μπροστά μας. Ελπίζω να τα καταφέρω μέχρι το τέλο τη θητεία. Ας δείξω κι εγώ πνεύμα αισιοδοξία, όπως η κυρία Ρέγνερ, αλλά πιστεύω ότι θα είναι πολύ περιπλοκό αυτό το πράγμα. Πολύ δύσκολο. Χρειάζεται υψηλή συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων, διαθεσμική καλή συνεργασία, για να μην χάσουμε την ουσία της πρότασης, το ψητό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για το θέμα των καταγγελόντων. Το ξέρατε το πρόβλημα και πριν. Το είπατε κι εσείς. Αλλά τα τελευταία, ε, τα χρόνια ε, και τους τελευταίους μήνες υπήρξε μια επιτάχυνση, ειδικά μετά τη δολοφονία στη Μάλτα. Σας ευχαριστώ για την ισορροπία του κειμένου, που, για το γεγονός ότι δεν μπερδεύεται το ρόλο ενός ε, καταγγέλλοντα, ενός πληροφοριοδότη με το ρόλο του δημοσιογράφου. Ε, πολύ συχνά στις συζητήσεις μας είχα την αίσθηση ότι μιλάμε για όλους, μπερδεύουμε τις πηγές του δημοσιογράφους και τους πληροφοριοδότες, σαν να είναι όλοι ένα πράγμα. Σαν να είναι όλοι πληροφοριοδότες. Το πακέτο για τους πληροφοριοδότες είναι πολύ ειδικό. Δεν είσαι καταγγέλων, εξ επαγγέλματος. Γίνεσαι όταν βλέπεις το χώρο εργασία σου, όταν βλέπεις την κοινότητά σου, όταν βλέπεις το περιβάλλον σου, κάτι το οποίο είναι λάθος Θέλεις να ενημερώσεις τότε τους άλλους. Και στην πρόταση οδηγία σας ε, αυτό που προτείνετε είναι πολύ σωστό. Το πλαίσιο είναι πολύ σωστό. Εάν εξειδικεύσουμε πολύ συγκεκριμένα τον όρο καταγγέλων, την ε, πηγή και το ποιος είναι δημοσιογράφος, ε, τότε δεν θα οδηγηθούμε σε λάθος συμπεράσματα και θα μπερδέψουμε τα πάντα. Αυτά για τους πληροφοριοδότες. Χθε μιλήσαμε με τον κύριο Τίμερ μας για το θέμα αυτό ενδελεχώς. Τώρα για το εταιρικό δίκαιο. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το θέμα του εταιρικού δικαίου και έχουμε προσπαθήσει και στο παρελθόν, αλλά, τα έχουμε, αλλά έχουμε αποτύχει. Ελπίζω αυτή τη φορά, παρότι έχουμε μπροστά μας μόνο ένα χρόνο πριν τελειώσει η θητεία μας, θα τα καταφέρουμε. Ελπίζω να Ασχοληθώ με την εφιλόδοξη αυτή πρόταση που παρουσίασε η, Επίτροπος, η Επιτροπή γενικά. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που τονίσατε στην παρουσίασή σας ότι η πρόταση θέλει να βοηθήσει τους τίμιους επιχειρηματίες. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αντιμετωπίζουμε τις ε, επιχειρήσεις σαν πιθανούς εγκληματίες, γενικά. Κάποιοι όντως έχουν ε, καταχραστεί το δίκαιο, ε, αλλά οι περισσότερες επιχειρήσεις αποτελούνται από τίμιους ανθρώπους, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι ο τομέας αυτός προσφέρει το 80% των θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πλειάδα τέτοιων επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο αριθμό των επιχειρήσεων. Εκεί στηρίζεται η ευρωπαϊκή οικονομία, όχι στις μεγάλες πολυεθνικές στηρίζεται στις μικρές εταιρείες, στηρίζεται στις μικρομεσαίες εταιρείες. Για αυτές πρέπει να κάνουμε προτάσεις, γιατί εκεί εργάζονται οι πολίτες μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να μας πείτε πώς θα τα καταφέρουμε να τελειώσουμε το θέμα αυτό μέχρι το τέλος αυτής της θητείας. Ή τουλάχιστον αν δεν τελειώσουμε, τουλάχιστον να προχωρήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Κυρία Ροζιέρ, σύντομα παρακαλώ για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, Επίτροπο που ήρθε και για την ε, πρόταση τη χτεσινή που βέβαια ανταποκρίνεται σε αυτό που έχουν ζητήσει οι σοσιαλδημοκράτες εδώ και καιρό για την προστασία των καταγγελόντων. Και χαιρόμαστε που υπάρχει κάποια εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί στην αρχή δεν φαινόταν τόσο προφανές να έχουμε ένα νομοθετικό κείμενο αλλά τελικά εισακούστηκε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίω αυτό των σοσιαλδημοκρατών και μας προτείνατε μια, ένα νομοθετικό κείμενο σύμφωνα με τα όσα έχει εγκρίνει εδώ και πέντε μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Είναι μια πρόταση η οποία καλύπτει σε ένα μεγάλο βαθμό τους τότε στόχους μας. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ που εισακούστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρχαν πολλά θέματα σε εκκρεμότητα για το πεδίο εφαρμογή, για παράδειγμα, που δεν περιορίζεται μόνο στους μισθωτούς, μόνο σε αυτή την εργασιακή σχέση, αλλά καλύπτει η πρόταση και πολλούς ε, τομείς αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το είχαμε ζητήσει, δηλαδή οριζόντια προστασία και όσο γίνεται περισσότερο ευρεία. Και αυτό το χαιρετίζουμε λοιπόν η νομική επίση συμπαράσταση, όλα αυτά πηγαίνουν προ τη σωστή κατεύθυνση και μπορείτε να βασιστείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ομάδα μα ιδιαίτερα για να υπάρξει και παρετέρω Το πεδίο εφαρμογή είπαμε ότι είναι αρκετά ευρύ, αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε ακόμα περισσότερο τα πράγματα για καταγγελίε οι οποίε δεν έχουν να κάνουν τόσο με παράνομα πράγματα. Το LuxLeaks, για παράδειγμα, είναι μια υπόθεση που μα συνόδεψε σε όλη αυτή τη θητεία. Οπότε εμεί και σε τέτοιε περιπτώσει θέλουμε προστασία. Πάντα για το πεδίο εφαρμογή. Ε, το θέμα του εργασιακού δικαίου δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει μια τέτοια προστασία. Και έχω και μια ερώτηση για την εφαρμογή συγκεκριμένα την υλοποίηση. Έχουμε λοιπόν νομικό πλαίσιο προστασία, εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα ποιοι είναι καταγγέλλοντες, είναι άτομα μόνα τους, απομονωμένα, που δεν έχουν συνομιλητή, δεν έχουν σε ποιον να απευθυνθούν, δεν πρόκειται για ομάδες. Αντίθετα, είναι από την άλλη μεριά των ομάδων που εκείνες έχουν ε, όλες τις δυνατότητες και τη δύναμη. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει θεσμικός συνομιλητής και ανεξάρτητες αρχές που να μπορούν να συνομιλούν με τους καταγγέλλοντες, να μην νιώθουν ε, μόνοι τους, να μην νιώθουν δυσκολία στο να βγούνε προς τα έξω. Τέλος, υπογραμμίσατε τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Πράγματι μπορείτε να βασιστείτε σε αυτήν. Οι Υπουργοί όμως τι λένε γι' αυτά. Θα προχωρήσουν γρήγορα οι χώρες μέλη. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις, κυρία Επίτροπε. Τώρα η πρόκληση που έχετε μπροστά σας, κύριε Επίτροπε, είναι να απαντήσετε στο λίγο χρόνο που μας μένει. Η Επίτροπος, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που λέτε, που όντως βοηθούν να διευρύνουμε και εμείς τη σκέψη μας. Λοιπόν, να απαντήσω σε μια ερώτηση που επαναλάβατε πολλές φορές για το χρονοδιάγραμμα. Και ο κύριος Σφίσκα ε, με ρώτησε πόσο σίγουρη είμαι. Εγώ μπορώ να είμαι σίγουρη μόνο για αυτό που θα κάνω εγώ. Εγώ θα πιέσω, γιατί άλλα δεν μπορώ να πω ότι είμαι σίγουρη. Εγώ θα πιώσω λοιπόν την Προεδρία και την επόμενη Προεδρία, το πρώτο εξώμενο της επόμενης χρονιάς, στη Ρουμανική, για να προχωρήσει. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους και για όλα, γιατί για τα, τις ψυχιακές συμβάσεις χρειάζεται χρόνος. Εγώ τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον ε, Βούλγαρο Υπουργό. Είχα ήδη δύο συναντήσεις μαζί του νωρίτερα, προκειμένου τον ε, πίσω, να πιέσει και αυτός περισσότερο για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουν αυτές οι υποθέσεις στον χρόνο. Υπό την Αυστριακή Προεδρία πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν. Ελπίζουμε τουλάχιστον. Όσον αφορά τις νέες πρωτοβουλίες τώρα, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Όσον αφορά τα θέματα αστικής δικαιοσύνης, είμαι ανήσυχη, γιατί υπάρχουν πολλές καλές προθέσεις αλλά έχουν να κάνουν και με τις λεπτομέρειες. Οπότε δεν σας κρύβω την απογοήτευσή μου όσον αφορά την πρόοδο. Στις Βρυξέλλες δεν προχωράμε πολύ για την ρύθμιση α. Στην αρχή όλοι είχαμε την ίδια άποψη ότι τα παιδιά δεν πρέπει να βρίσκονται σε δύσκολη θέση μετά το διαζύγιο των γονιών τους Έχουμε να κάνουμε όμως εδώ με τις λεπτομέρειες. Σε αυτές κολλάμε. Υπάρχουν καλές προθέσεις, αλλά όπως ξέρουμε, συχνά οι καλές προθέσεις οδηγούν στην κόλαση. Τέλος πάντων, συγγνώμη που σας το λέω αυτό. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό εδώ. Η συλλογική αποζημίωση πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει αλλά είναι ακόμα θέματα αρμοδιότητα που μας προβληματίζουν, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και χωρών μελών, και για την αφαιρεγκαιότητα και για τους καταγγέλλοντε. Τώρα θα αρχίσω με τους καταγγέλλοντες, γιατί πολλά με ρωτήσατε γι' αυτό και υπήρξαν και πολλά σχόλια. Και πώς αποφασίσαμε για το ε, πεδίο εφαρμογής που μπορεί να υπάρξει μεγάλη ζημιά για το κοινό. Αυτό ήταν ο ένας πυλώνας, ο βασικός. Και ο άλλος ήταν να προστατεύσουμε τους τίμιους ανθρώπους, να τους ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσουν τις διόδους που έχουν στη διάθεσή τους Στι διαπραγματεύσει, πιθανόν να διαβρεθεί ακόμα περισσότερο το πεδίο εφαρμογή. Προ το παρόν πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν βλέπει τις δυνατότητε γιατί η νομική βάση είναι η ενιαία αγορά και τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελέγξαμε όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να προκύψει μεγάλη ζημιά για το κοινό. Τώρα στις διαπραγματεύσεις μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο το πεδίο εφαρμογή και ίσως να υπάρξουν νέες ιδέες που θα ευθυγραμμίζονται όμως με την νομική βάση έτσι, για την προστασία αυτή των καταγγελόντων, τη σχετική οδηγία. Με διέφερε πάρα πολύ η νομοθεσία αυτή. Δεν ήθελα να φτάσουμε σε κάτι που θα είναι η προστασία των καταγγελόντων ή για την προστασία των καταγγελόντων. Εμένα με ενδιαφέρει η προστασία του κοινού. Γι' αυτό και λάβαμε υπόψη μας όλες τις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρξει τέτοια ζημιά. Επνευστήκαμε και από τα LuxLeaks και από την περίπτωση του Cambridge Analytica πρόσφατα. Και γι' αυτό καταλήξαμε να λάβουμε υπόψη μας ε, τους κινδύνους για σοβαρή ζημιά. Ε, για το χρονοδιάγραμμα πάντα, όσο γίνεται πιο γρήγορα θα μιλήσω με την Βουλγαρική Προεδρία για να πιέσουμε. Και την πρόταση όσον αφορά τους καταγγέλλοντες και τη Μάλτα, ναι, θα έρθω στο θέμα της Μάλτας και υπάρχουν πολλά που πρέπει να καλύψουμε εκεί όπως επίσης η καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομου χρήματος. Υπάρχουν τα θέματα που έχουν να κάνουν ε, με τις ε, πληροφορίες όσον αφορά το φαινόμενο αυτό. Οπότε θα ζητήσω να μάθω από τη Μάλτα τι συγκεκριμένα μέτρα παίρνει. Και θα ζητήσω και από την εισαγγελία να ξέρω πώς προχωράει η έρευνα όσον αφορά τον ε, θάνατο της δημοσιογράφου Αυτά βέβαια συνδέονται με τους καταγγέλλοντες και με την προστασία των δημοσιογράφων. Γιατί σύμφωνα με τον νόμο βέβαια, οι δημοσιογράφοι δεν εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή της προστασίας καταγγελόντων, γιατί έχουν προστασία σε εθνικό επίπεδο. Η δικιά μας όμως οδηγία αυτή για τους καταγγέλλοντες σίγουρα θα τους βοηθήσει, γιατί αν μη τι άλλο οι πληφοριοδότες τους, οι πηγές τους, θα έχουν ε, λιγότερους δισταγμούς να πάνε στους δημοσιογράφους και να μιλήσουν με αυτούς. Θα νιώθουν ότι έχουν προστασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να ξεπερνάει τους δισταγμούς τους. Εδώ δεν πρόκειται για τη δημοσιογραφία, αλλά ξέρετε υπάρχει και η ρητορική μίσους. Και εδώ έχουμε την αυτολογοκρισία. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι όλο και περισσότερο ανταλαμβάνονται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο. Υπάρχουν απειλές online, υπάρχουν μερικά πολύ σκληρά μηνύματα. Οι χώρες μέλη πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτό και να φροντίσουν για την προστασία των δημοσιογράφων. Είναι θέμα χωρών μελών πάντως και όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η απάντησή μου και σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Καβαντά για την προστασία των δημοσιογράφων. Και για το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας για τους καταγγέλλοντες. Για τη Μάλτα πάλι δεν έχουμε στοιχεία για ανάμιξη του κράτους της Μάλτας. Πιέζουμε όμως για να έχουμε τα αποτελέσματα όλων των ερευνών και ανακρίσεων που γίνονται στη Μάλτα. Γι' αυτό και θέλω να πάω στη χώρα και να συναντηθώ με τους υπεύθυνου και να τους ρωτήσω γι' αυτό. Πολλά ήταν για τους καταγγέλλοντες. Η απόφαση καπιτάνη. Δουλεύουμε πάνω στη νομική θέση και ακολουθούμε βεβαίως την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λέει κυρία Γιούροβα. Κύριε Ροζιέ, Ναι, λέτε ότι εισακουστήκατε. Εντάξει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πάντα προσπαθούμε να ακούμε τι λέτε. Για την προστασία των καταγγελόντων υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό που πρέπει να πω όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή και τα LuxLeaks. Ο καταγγέλων, ο οποίος ανακοίνωσε, μίλησε για την φόρο αποφυγή, τιμωρήθηκε. Αυτό λοιπόν που εμείς προτείνουμε εδώ είναι ότι δεν θέλουμε να υπάρξει διαφοροποίηση αν κάνει κάτι παράνομο. Όμως, αν δεν κάνει κάτι παράνομο και τίμια ανακοινώνει κάτι, δεν πρέπει να τιμωρείται άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, τα LuxLeaks είναι μια καλή περίπτωση που δείχνει γιατί προτείνουμε το κείμενο όπως το προτείνουμε. Ανοίγουμε εσωτερικές διόδους για καταγγελίες και πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών να ενημερώνεται ο κόσμος για την ύπαρξη αυτών των εσωτερικών ε, καναλιών ώστε να ξέρει ο κόσμος ότι αν καταγγέλει κάτι είναι προς το συμφέρον της καλής διαχείρισης του οργανισμού για τον οποίο υπάρχει καταγγελία. Αν δεν λειτουργήσει η εσωτερική δίωδος, έχουν εξωτερική αντίστοιχη. Και πρέπει να είναι ενημερωμένος ο κόσμος, να ξέρει πού πρέπει να πάει για να αναφέρει μια καταγγελία. Και θα πρέπει λοιπόν η ενημέρωση αυτή να γίνεται σε όλες τις χώρες, να ξέρει ο κόσμος που πρέπει να απευθυνθεί. Εμείς δεν λέμε αν πρέπει να είναι ένα κεντρικό σώμα ή τομεακά σώματα. Μπορεί να χρειαζόμαστε περισσότερα του ενός οργάνου για τέτοιες καταγγελίες. Αλλά το βέβαιο είναι ότι παντού και πάντα πρέπει να ξέρουν οι καταγγέλλοντες ότι έχουν που να απευθυνθούν. Και έτσι κι αλλιώς υπάρχει πάντα ο συνήγορος του πολίτη, στον οποίο μπορεί να απευθυνθεί. Και αν τέλος πάντων δεν έχει λειτουργήσει τίποτα από τα δύο πρώτα στάδια, τότε θα πρέπει οι καταγγέλλοντες να βγαίνουν στον τύπο, στο κοινό, και θα πρέπει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και τις τρεις να υπάρχει η ίδια προστασία των καταγγελόντων. Αλλά πρώτα απ' όλα ενημέρωση, να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί που μπορούν να απευθυνθούν. Τώρα για το επιχειρηματικό δίκαιο. Ναι, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικό στοιχείο εδώ. Είναι ένα πακέτο, όντως ε, αργήσαμε περισσότερο από το αναμενόμενο. Πρέπει όμως να παραδεχτώ ότι άλλαξε η υπόθεση και με την απόφαση του δικαστηρίου. Οπότε θέλαμε να έχουμε μια νομοθεσία που να επιτρέπει την διασυνοριακή μετακίνηση των επιχειρήσεων, αλλά η δικαστική αυτή απόφαση έχει μια πιο πώς το αντιμετώπιση και έπρεπε έτσι να ξαναδούμε ολόκληρο το πακέτο μετά την απόφαση αυτή και να έχουμε περισσότερες ρήτρες ασφάλειας για ενδεχόμενες καταχρήσεις. Και εδώ είναι που το πακέτο συνάδει με τις ιδέες για την κοινωνική Ευρώπη του Ζανκλώτ Γιούγκερ, γιατί προβλέπει την συμμετοχή των καταναλωτών και εμείς συμφωνούμε εφόσον υπάρχει στη χώρα μέλος πρέπει να τηρείται και στη διαδικασία. Γι' αυτό και έχουμε διατάξεις κατά των επιχειρήσεων θηρίδων και κατά των καταχρήσεων των διασυνοριακών μετακινήσεων που θα έβλεπταν τους μετόχους ή τους ε, εργαζόμενους. Θα τα δείτε όλα αυτά, θα τις δείτε όλες αυτές τις δικλίδες ε, ασφαλείας. Θέλω να προστατεύσω τους τίμιους επιχειρηματίες βέβαια, αλλά ήταν αναγκαίο να υπάρχουν αυτές οι κλίδες ασφαλείας για να προστατεύσουμε τον κόσμο από καταχρήσεις. Και συμφωνώ με τον κύριο Ζιέφκα πλήρω. Πολύ θα ήθελα κι εγώ η νομοθεσία να γίνεται για τους τίμιους ανθρώπους. Και αυτό έγινε και με την αφαιρεγκαιότητα. Άκουσα τις φωνές κατά των καταχρήσεων. Άκουσα αυτούς που λένε ότι η ψηφιοποίηση του επιχειρηματικού δικαίου είναι η λύση για να μην υπάρχουν καταχρήσεις, καταχώρηση online, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να ελέγξει τα γεγονότα αν όντως ιδρύθηκε μια εταιρεία. Ό,τι και αν κάνουμε, προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί. Για μένα προτεραιότητα έχει η πεποίθηση ότι η νομοθεσία μας πρέπει να εξυπηρετεί τους τίμιους επιχειρηματίες. Για τις συμβιακές συμβάσεις, όπως είπα και πριν, πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε την ε, έγκριση πακέτου. Μπορώ σήμερα να επιβεβαιώσω ότι δεν θέλω να μειώσω το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε οποιαδήποτε χώρα μέλος. Πρέπει να βρούμε διέξοδο ήταν και ερώτηση της κυρίας Χαουτάλα. Δεν θέλω να μείνω γνωστή σαν την Επίτροπο Προστασίας των Καταναλωτών, που μείωσε όμως το επίπεδο προστασίας στην Ιρλανδία ή στη Φιλανδία, έξω που. Όχι, πρέπει να υπάρξει αναρμόνιση των κανόνων και να επιτρέψουμε στις χώρες μέλη που θέλουν μεγαλύτερη προστασία να μπορούν να την έχουν να μπορεί κανείς να ανεβάσει το επίπεδο προστασίας εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο επίσης και για το ενσωματωμένο software. Και αυτό πρέπει να γίνει για το μέλλον. Να καλύψουμε και το διαδίκτυο των πραγμάτων, γιατί όλο και περισσότερο τα κουτιά θα είναι το σημαντικό. Να ξέρουμε ποιοι μπορεί να είναι οι επικίνδυνοι, οι, επόμενοι κίνδυνοι για τους καταναλωτές. Εγώ θέλω απλοποίηση, απλούστευση. Δεν μπορούμε στους καταναλωτές να προσφέρουμε κάτι περίπλοκο που θα οδηγήσει σε διαφορετικά καθεστώτα για το software, για τα κουτιά, για τις υπηρεσίες κτλ. Δεν το θέλουμε αυτό. Γι' αυτό εδώ πρέπει να βρούμε λύση. Κύριε Ντελβό, ναι, ρομποτική. Ξέρω ότι περιμένετε περισσότερα, αλλά θα έχουμε την πρότασή μας περί και ασφάλειας του χρόνου. Προς το παρόν, η πρότασή μας, η ανακοίνωση που θα εγκρίνουμε αύριο, θα καλύπτει τη στήριξη της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει εφιούς χρηματοδότησης και στήριξης της έρευνας. Νωρίτερα ολοκλήρωσα την ομιλία μου λέγοντας ότι μπορούμε να είμαστε σε ηγετικό ρόλο, αλλά είναι δύσκολο γιατί έχουμε την Κίνα, έχουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες, οι οποίες τι κάνουν, μαζεύουν τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων χωρίς δισταγμούς. Δεν σέβονται την ιδιωτικότητα των ανθρώπων. Είδατε τι έγινε με την ε, Cambridge Analytica και το Facebook. Δεν σέβονται το άτομο. Γι' αυτό και θέλουμε εμείς τα δεδομένα να μπορούμε να τα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα τα δικαιώματα των ατόμων. Θα το κάνουμε έτσι όπως ξέρουμε να το κάνουμε εμείς στην Ευρώπη. Με έρευνα που θα πηγαίνει χέρι-χέρι με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα το κάνουμε με τον ευρωπαϊκό τρόπο και είμαι σίγουρη ότι θα πετύχουμε. Γι' αυτό λοιπόν η αυριανή μας ε, πρόταση θα αφορά την έρευνα, την ευφύ χρηματοδότηση και την ανάγκη να προστατέψουμε τα συστήματα εκπαίδευσης ώστε να υπάρχει προσαρμογή στη νέα αγορά. Και κατά τη γνώμη μου έτσι θα ερμηνεύσουμε καλύτερα και το σημερινό νομικό πλαίσιο. Θα δούμε δηλαδή πώς πρέπει να το εφαρμόζουμε σε περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν και να έχουν να κάνουν με θέματα περί Η ερμηνεία μας είναι ότι οι γενικοί κανόνες για την ασφάλεια των ε, προϊόντων θα ισχύσει και εκείνη για τις μηχανές και του χρόνου θα έχουμε και σύσταση προκειμένου να συνεχίσει πάνω σε αυτήν η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για νέα νομοθεσία. Στην εντολή μας πάντως θα κάνουμε ακόμα πολύ αναλυτική δουλειά για να την προσφέρουμε στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπου δεν χρειάζεται νέα νομοθεσία, ας ισχύσουν και σε εφαρμοστούν καλύτερα οι σημερινοί κανόνες περί ευθύνες. Αυτό θέλουμε για του χρόνου. Και... Έντουαρτ, ναι, έχετε δίκιο. Θα ολοκληρώσω εδώ πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλές σας ερωτήσεις και τα σχόλια. Η κυρία Χατάλα, κύριε Επίτροπε, μπορείτε έστω και σύντομα να απαντήσετε στην ερώτησή μου όσον αφορά την πρόσφαση στη δικαιοσύνη εκείνων που είναι θύματα ε, επιχειρηματικών συνασπισμών. Υπάρχει αυτό που σας είπα προηγουμένως για τις ε, διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Γιατί το πεδίο εφαρμογή για τη συλλογική αγωγή που προτείνουμε, όπως ξέρετε, ήταν πολύ στροπημένο. Το είχαμε σκεφτεί πολύ καλά. Και έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις, σας διαβεβαίω, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, στην αρχή πρέπει να σας ομολογήσω ότι ήμουν απογοητευμένη, γιατί ε, από ό,τι φαινόταν θα καλύπταμε ένα πολύ περιορισμένο κομμάτι της προστασίας των καταναλωτών. Στη συνέχεια, οι συνάδελφοι δεν μπορούν να πω ότι ξύπνησαν, δεν κοιμόντουσαν ποτέ, αλλά όλο και πιο πολύ υπέβαλαν ιδέες για τη συλλογική αγωγή που θα κάλυπτε και τους δικούς τους τομείς αρμοδιότητας ενδεχομένω στι διαπραγματεύσει ε, να κάνετε προτάσει εσεί ή να γίνουν προτάσει από πλευρά των κρατών μελών. Εμά το σκεπτικό μα ποιο ήταν να προβλέψουμε πού μπορεί να προκληθεί μαζική ζημία. Και που οι συλλογικές αγωγές θα αποτέλεσαν το κατεξοχήν ε, πλέον κατάλληλο εργαλείο για τη μετώπιση των ζητημάτων αυτών. Αν ε, βρείτε και άλλα θέματα που θέλετε να καλυφθούν, ε, αυτό θα αποτελέσει έργο των συνομοθετών. Αλλά εμείς προσβλέπουμε στη συζήτηση. Ευχαριστούμε, Επίτροπε Γιούροβα, για την ανταλλαγή αυτή απόψεων που πραγματικά μας εμπλουτίζουν. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εμένα με εμπλουτίζουν. Σας ευχαριστούμε και προσβλέπουμε λοιπόν και την επόμενη φορά που θα έρθετε στην Επιτροπή μας. Dear colleagues, uh, are prepared... Συνάδελφοι, είμαστε έτοιμοι για ψηφορίες. Δεν είναι όλοι τιμή μου φαίνεται. Μάλιστα να ψηφίσουμε για το σχέδιο της έκτασης του προπολογισμού του το 2016 το σχετικό σκόρμπορ, το πίνακα των αποτελεσμάτων. Πρώτον το θέμα αυτό, στον τομέα της δικαιοσύνης. Συμβιβαστική Β, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Λίμπα Οκτώ. υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται. Λείπε 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λείπε 14. Τη λείπει 8, θέλετε να ελέγξουμε. I did say, I did say Είπα ότι απορρίφθηκε. Αν θέλετε να το ελέγξουμε, το ελέγχουμε πάντως. Βεβαίως. Ηλεκτρονικός έλεγχος. One more. Μία ψήφος ακόμα. Πολύ ωραία. Εγκρίθηκε. Ζητώ συγγνώμη. Λίμπε 14, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική M, υπέρ. Κατά. Άποχες Εγκρίνεται. Λίπε 16. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Σεμιβαστική σί, Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται ή 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική G. Υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται η 57 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται συμβαστική ήττα H υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται συμβαστική I Ι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ για την 71 ηλεκτρονικός έλεγχος απορρίφθηκε 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ για την 88. Εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 90. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική α υπέρ κατά Απόχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 και 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ για την 17 ε, και 19 ταυτόσημες. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Η 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ ηλεκτρονικός για την 1. Άλλη μία ψήφος. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 και 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος, ε, γιατί νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά δεν είμαι και βέβαιος. Για την τρία παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος. Εγκρίθηκε. Και τώρα ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης. Και πέρα της ψηφορίας εγκρίθηκε και συγχαρητήρια στην κυρία Γκούτλαντ. Και τώρα να ψηφίσουμε το σχέδιο έκθεση για την αντικατάσταση του παρακτήματος Α του κανονισμού 2015-848 περί των διαδικασιών αφαιρεγγιότητας. έχουμε μία ψηφοφορία αμπλόκα ε, για όλες τις τροπολογίες. Θέλετε να το κάνουμε ηλεκτρονικά. Για να απολαύσουμε πιο πολύ τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Άλλε δύο ψήφοι και τώρα ολοκληρώθηκε λοιπόν ο κατάλογος και εγκρίνεται το σύνολο. Και τώρα το σχέδιο της έκτασης, το σύνολό του και πάλι ηλεκτρονικά όμως. Μεγάλη έκπληξη, μεγάλη αγωνία. Εγκρίθηκε και συγχαρητήρια προς τον κύριο σε Συγχαρητήρια. Τώρα, Περνάμε στις στατιστικέ σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω ιστορικών πλουτών οδών, κωδικοποιημένο κείμενο, ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε παρακαλώ, έναρξη τη πληροφορία. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια την κυρία Γκέρινγκερ. πρότυπα επιδόσεων για τι εκπομπές. Ηλεκτρονικά και πάλι ψηφίζουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε και πάλι συγχαρητήρια στην κυρία Γκέρνιερ. Αυτά και έτσι ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες σήμερα. So, no. Yes. Yes. Και τώρα θα θέλαμε να συνεχίσουμε με το σημείο 6 της ημερής να ανακοινώσει του Πρόεδρου. Καταρχάς, να σας πω ότι η κοινή σε Γιούρι και Αύκο με ψηφοφορία για το σχέδιο της έκθεσης για την εφαρμογή και την ερμηνεία της, καλύτερης, της Συμφωνίας Καλύτερης Νομοθεσίας θα λάβει χώρα αύριο στις 11.50. 11.50, τονίζω. 12 παρά 10. Πολύ ωραία. Κατά δεύτερον, η συνάντηση για το Brexit με το Υπουργείο Ιστορικών του Ηνωμένου Βασιλείου θα λάβει χώρα σήμερα στις 12.30 στην αίθουσα ASP 5G3 μετά την πρωινή μας συνεδρίαση. η Επιτροπή Γιούρι έχει προσκληθεί στην συνάντηση αυτή. Στη συνέχεια να σας ενημερώσω για την απόφαση των συντονιστών χτες το βράδυ. Οι συντονιστές λοιπόν συμφώνησαν να ορίσουν την κυρία Χάουτελα για την έκθεση για την άρση της ε, ασυλίας του κυρίου Γιώργιου Κίτσου. Να ορίσουν τον κύριο Σβιεύκα εισηγητή για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την ε, ε, ταχεία επεξεργασία διαφωνιών, τον κύριο Μάσταλκ για τους εργαζομένους και τους κινδύνους από καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνε ουσίες στην δουλειά και σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και την βιωσιμότητα της ε, αξιολόγησης των τροφίμων και της αλυσίδας των τροφίμων και ύστερα η οδηγία για την ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων. Να καλέσουμε τον Επίτροπο Ότιγκερ Αποφασίσαμε να συμμετέχει στο διαρθωμένο διάλογο με την Επιτροπή και να, σύνουμε, να στείλουμε επίστολη σε αυτόν σε ό,τι αφορά το υψηλό προσωπικό και να επιστήσουμε την προσοχή του στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Γιούρη σε ό,τι αφορά θέματα κανονισμού α, για το ιστορικό κανονισμού και να αποσταλεί σχετική επιστολή στον επικεφαλής της Επιτροπής Και τέλος, οι, οι συντονιστές αποφάσισαν να γίνει μια ανεπίσημη συνάντηση με τον α, συντονιστή για θέματα πραγματικών δικαιωμάτων από πλευρά των ΗΠΑ. Αυτές λοιπόν ήταν οι ανακοινώσεις μου. Now we are at item 7. Πάμε στο σημείο 17. Καλωσορίζουμε τον απερχόμενο εκτελεστικό διευθυντή του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριο Αντώνιο Καμπίνος, για να μιλήσει για μια τελευταία φορά στην Επιτροπή μας, ως, με την ιδιότητά του του εκτελεστικού διευθυντή, πριν αναλάβει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Γραφείου ε, Ευρεσιτεχνιών πρώτης 1η Εβδόμου του 2018. Συγχαίρω για τον νέο σου this... Ο σκοπός της ανταλλαγής να συζητήσουμε τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Γραφείου, ε, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έχει. Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια ήσασταν πολύ ε, ε, γενναιόδοροι, με το χρόνο σας ε, και δώσατε μεγάλη σημασία στα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Είμαστε ευγνώμονες για την προσοχή και για τις προσπάθειες που κάναν τα μέλη της Επιτροπής για να υποστηρίξουν την βελτίωση στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προς το συμφέρον των χριστών και των Ευρωπαίων πολιτών. Η εξελίξη τα τελευταία χρόνια ε, και η πίεση των τελευταίων γεγονότων έδειξαν ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, ενδιαφέρεται πολύ για την καινοτομία και για τη δημιουργικότητα και ήταν πραγματικά πρωτοπόρα. Ορισμένοι από εσά ξέρετε ότι είναι η τελευταία μου ευκαιρία να μιλήσω στην Επιτροπή σα ω εκπαιδευτικό διευθυντή του Γραφείου Διανοητική Ιδιοκτησία, μια και είπε ο Πρόεδρο ότι από πρώτη εβδόμου θα πάρω ε, τη θέση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Γραφείου ε, Ευρεσιτεχνιών. Με ενδιαφέρει η δημιουργικότητα, η καινοτομία και κυρίως η εφεύρεση. Ε, καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο ε, σκέφτομαι και τη διασύνδεση ανάμεσα στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και την ανάγκη για μια κοινή προσέγγιση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίω για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να υποφεληθώ από την ευκαιρία να υπενθυμίσω κάποιες από τις αλλαγές που έχουν ήδη λάβει χώρα ε, στο πεδίο της διανοητικής ιδιοκτησίας και να σας μιλήσω για τις ε, μελλοντικέ προκλήσεις, οι οποίες ε, αφορούν το, τη γρήγορη τεχνολογική αλλαγή, την τεράστια ζήτηση για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας παγκόσμια και πώς θα εξασφαλίσουμε ότι γίνονται σεβαστά στην παγκόσμια αγορά θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή 7 και πλέον χρόνια πίσω ε, από την πρώτη φορά που μίλησα στην Επιτροπή σας το 2011, από την πρώτη ε, συνάντηση, ε, μέσα σε ένα χρόνο από τότε, η διανοητική διοκτησία αυξάνεται σε σημασία πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά. Οι ευθύνε του γραφείου εξελίσσονται φυσικά αντίστοιχα. Το γραφείο ε, συνεισφέρει τώρα σε όλους τους τομείς ε, δικαιωμάτων γενετικής ιδιοκτησίας, όχι ως γραφείο καταχώρησης ε, ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων και σχεδίων. Ορισμένοι ε, λένε ότι πραγματικά παίζουμε το ρόλο ενός γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας 100%. Και αυτό δεν θα είχε γίνει χωρί την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Κομισιόν και του Συμβουλίου και την υποστήριξη όλων των ενδιαφερομένων καθώς και των ε, χρηστών του συστήματος ε, δικαιωμάτων που έχουν γίνει εταίροι σε αυτήν την προσπάθεια. Το 2011 είχα μιλήσει για τη σημασία των δικαιωμάτων αυτών για την οικονομία και την κοινωνία εν γέννη. Από τότε το γραφείο ασχολήθηκε ε, και ενισχύθηκε από το παρατηρητήριο με, που ασχολείται με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων το 2012 και μετά από 40 μελέτες για το ρόλο του, ε, τη διανοτική ιδιοκτησία ιδιοκτησίας στη μοντέρνα κοινωνία, τα θέματα αυτά έχουν ξεκαθαριστεί περισσότερο. Οι οικονομικές κυρίως μελέτες για τη σημασία των δικαιωμάτων, οι βλάβες από τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων και την αντίληψη που έχουν οι πολίτες για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας είναι, αποτελούν ένα τρίγωνο. Και τώρα τα δέχονται παγκοσμίω και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς. Οι μελέτες παρατέθηκαν ε, από πολλούς, ε, από το G7, ε, ακόμα και τον, από τον ΠΟΕ στη Γενέβη πρόσφατα, όπου η Κομισιόν εκλήθη για να παρουσιάσει το έργο της για την επίπτωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ε, στην οικονομία ε, στο Συμβούλιο TRIPS. Ο τρίλογος, το τρίγωνο αυτό επικαιροποιείται και συμπληρώνεται από πολλές εξετάσεις που καλύπτουν το χαμένο δυναμικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τι μπορούμε να κάνουμε για να καλύψουμε αυτό κενό. Για να το κάνουμε αυτό, έχουμε μια πιο στενή εταιρική σχέση με άλλα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας και φορείς ε, στα πλαίσια της διαδικασίας ε, της ψηφιοποίησης ε, των εμπορικών σημάτων και σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μειώσουμε το κόστος αλληλεπίδρασης με πολλές ε, άλλες υπηρεσίες για να προστατεύσουμε τα διανοητικά δικαιώματα, ε, έχουμε 7 πεδία σύγκλησης, ε, δύο από αυτά καλύπτουν τα σχέδια. Υπάρχουν και άλλα σχέδια σύγκλησης που αφορούν θέματα εμπορικών σχεδίων και αποκάλυψης των σχεδίων στο ίντερνετ. Στο Επίσης, τι γίνεται με, την ε, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, που είναι σημαντικός αν θέλουμε να υποφελθούμε από την καινοτομία ε, και τη δημιουργικότητα. Ε, σας επιβεβαιώνω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι εταιρικέ σχέσεις συνεχίζονται και επεκτείνονται και σε άλλα διανοητικά δικαιώματα, καθώς και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Είναι πολύ βασικό για να εποφεληθούμε από το δυναμικό που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτω ώστε οι εφευρέσεις να γίνουν εμπορικά προϊόντα. Ε, μιλάμε και για τις συμφωνίες αδειοδότησης που θα πρέπει να αναγνωρίζονται. Το γραφείο πρόσφατα κοίταξε τι μπορούμε να κάνουμε για να ενθαρρύνουμε την, ε, τη μεταφορά τεχνο, τεχνολογίας. Υπάρχει και μια πρωτοβουλία για να δημιουργήσουμε μια δικτυακή πύλη που θα μπορούσε να ε, λειτουργήσει ως ενιαία θηρίδα για εταιρείε που αναζητούν πληροφορίε για να τι βοηθήσουμε πώ να εκμεταλλευτούν τα δικαιώματα κοινωνική ιδιοκτησία. Το γραφείο συνεργάζεται σε δίκτυο ε, όλων που αποκαλύπτουν όλο το φάσμα των διανοητικών δικαιωμάτων. Ε, και το πιο σημαντικό, το πώ μπορούμε να τα καταλάβουμε καλύτερα αυτά τα δικαιώματα και να τα εφαρμόσουμε και να γίνουν σεβαστά. Υπάρχουν δραστηριότητε αφύπνιση του κοινού. Ε, συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικέ αρχέ, ούτω ώστε να υπάρχει και εκπαιδευτικό υλικό για τα διανοητικά δικαιώματα ε, στην εκπαίδευση. Θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε τις αρχές εφαρμογής ε, να υπάρχουν, ε, υπάρχει καλύτερη συνεργασία με δικαστές, με εισαγγε, τους εισαγγελείς και με την αστυνομία. Η πολύ σημαντική σχέση που έχουμε αναπτύξει επίσης με την Europol είναι σημαντική, όπου υποστηρίζουμε ένα κέντρο για τα δικαιωματικά δικαιώματα που υπάρχει για να καταπολεμήσουμε τα εγκλήματα παραβίασης δικαιωμάτων ιατρικής ιδιοκτησίας στο ίντερνετ. Ασχολούμαστε δηλαδή με όλο το φάσμα δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία. Συνεχίζουμε να εκπροσωπούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω φορέα εφαρμογή για διάφορα προγράμματα χρηματοδότηση σε πολλέ ε, περιοχές, ούτως ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκληση, μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη προσπελασιμότητα προ το συμφέρον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κυρίω. Ε, κάποιες από τι αλλαγέ που έγιναν στην κοινωνία και, στην και στο και στην οικονομία, τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Γι' αυτό κάναμε και νομοθετικές αλλαγές. Παρότι μπορούμε να πούμε ότι η νομοθεσία συχνά υπολείπεται σε σχέση με τις αλλαγές που γίνονται στην κοινωνία και στην οικονομία. Θα γνωρίζετε τις σημαντικές αλλαγές που έχουν κάνει στον οργανισμό για τα εμπορικά σήματα που οδηγεί σε απλούστευση, σε διευκρίνηση, σε διευκρινήσεις και διευκρινήσει και θέματα διεθνούς συνεργασία. Καθώ και τι επίσημε αρμοδιότητες του γραφείου. Τον Οκτώβριο πέρυσι ε, Υπάρχει και αίτημα για γραφική αποτύπωση των εμπορικών σημάτων, αλλά αυτό έχει καταργηθεί. Ε, οι χρήστες και εγώ πιστεύω και κάποιοι νομοθετές ζητούν να γίνει αντίστοιχη νομοθετική αλλαγή και στα σχέδια. Ευτυχώς το γραφείο καταλαβαίνει ότι ένα νέο κανονισμό για, τα σχέδια είναι κάτι που δεν θα γίνει άμεσα. Ε, παράλληλα, Υπάρχει παγκόσμια οικονομία σήμερα. Ε, μην ξεχνάμε ότι αλλού, ε, στην Νότια Κορέα, υπάρχει εξυγχρονισμός ε, των σχεδίων. Ε, Μπορεί να καταχωρήσει κανείς ένα σχέδιο, αυτό το κάνει στην Κορέα, αλλά όχι σε εμά, στην Νότια Κορέα. Ε, όλα αυτά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ε, και οι, ε, ε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας κτλ. είναι αλληλένδετα. Και αυτό θα πρέπει να αναγνωριστεί. Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήταγε από το γραφείο να ε, αναλάβει ε, αρμοδιότητες και για γεωγραφικές ενδείξεις. Ε, προς το παρόν όμως δεν έχουν γίνει συγκεκριμένες προτάσεις. Ε, Αρχίζουμε να συνεργαζόμαστε πιο στενά όμως με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για να εξετάσουμε τα γεωργικά, ε, τους γεωγραφικές, ε, τις αγροτικές γεωγραφικές ενδείξεις. Ούτως ώστε στο μέλλον να αναλάβουμε δράση. Ε, δίνω μεγάλη σημασία στα σχέδια και σας είπα ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πιο ε, γενικό και ενιαίο πλαίσιο για τα, τις γεωγραφικές ενδείξεις η Κομισιόν θα πρέπει να, το, να ασχοληθεί με το θέμα μόλις το επιτρέψει το πρόγραμμα εργασίας της. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να σας αναφέρω για τις δραστηριότητε του γραφείου είναι ότι είναι σημαντικό να ε, κάνουμε αυτό που πρέπει ως γραφείο καταχώρησης. Ε, ο ρόλος του γραφείου έχει επεκταθεί. Παρ' όλα αυτά δεν ξεχνάει ότι θα πρέπει να χορηγούμε το ε, εμπορικό, ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα με ένα αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή για μας. Ε, οι επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει ε, σε προχωρημένη τεχνολογική, ε, ψηφιακή τεχνολογία και σε διάφορες πρακτικές ε, έχουν επιτρέψει να εργαστούμε καλά μέχρι το 2017. Παρ' όλα αυτά, ε, ο όγκος των εργασιών για τα για την καταχώρηση των σημάτων, των εμπορικών σημάτων και των σχεδίων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Οι αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ βαθιές. Χάρη όμως στην ομαδική δουλειά και στην υποστήριξη ε, που έχουμε λάβει ε, και χάρη και στην τεχνολογία μπορούσαμε να εργαστούμε πιο αποτελεσματικά. Ε, θα συνεχίσουμε να δίνουμε ποιοτικέ υπηρεσίες στο εγγύς μέλλον. Θα ήθελα να σας αναφέρω και ένα-δυο στατιστικές. Πέρυσι τα, οι αιτήσει για τα εμπορικά σήματα ήταν ε, το βασικό μας έργο και ήταν ε, πολύ σημαντικό για τη χρηματοδότηση των εργασιών μας. Ε, η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 8%. Παρά την μεγάλη ζήτηση, νέα πρότυπα για τη δημοσίευση των εμπορικών σημάτων έγιναν και καταφέραμε να δώσουμε τις αποφάσεις εγκαίρως. Το 2017 είχαμε κέρδη λόγω αποτελεσματικής εργασίας ε, ύψους 5,9%. Ε, θέλω να τιμήσω το προσωπικό ε, το οποίο προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις, ε, δείχνει ζήλο και θέλει να κάνει ό,τι μπορεί για να αυξήσει την προσθέμενη αξία του γραφείου. Αυτές οι στατιστικές θα δίνουν μια γεύση για το ταξίδι που έχει κάνει το γραφείο υπό διαφορετικές, ε, διαφορετικά προγράμματα εργασίας για να γίνουμε πιο ευέλικτος οργανισμός ε, εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα διανοτικής ιδιοκτησίας. Ελπίζω ότι για σας οι αλλαγές αυτές ε, θεωρούνται προς την κατεύθυνση. Όπως ξέρετε, Όμω οι προκλήσει για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησία αυξάνονται. Τα τελευταία χρόνια ε, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020 να υποστηρίξει την ε, δημιουργικότητα για μια έξυπνη, ε, χωρίς χωρί αποκλεισμού, ανάπτυξη. Το 2020 είναι πρώτον πυλών. Αντιμετωπίζουμε την Ευρώπη χωρί το Ηνωμένο Βασίλειο και υπάρχει και η επίπτωση των τεχνολογικών ε, αλλαγών ε, και κάποια όρια ε, των, των νομοθετών για να αντιδράσουν. Μιλάμε για φοβερές τεχνολογικές αλλαγές, τεχνο, ε, το bitcoin, τα κρυπτονομίσματα, την τεχνολογία του blockchain, Ορισμένα πράγματα είναι συνα, συναφή για τα, προς τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. αλλά τα δικαιώματα ε, σχεδίου ε, έχουν μεγάλη σχέση για το τελικό προϊόν. Ε, υπάρχει δυνατότητα ε, ε με λέιζερ. Υπάρχουν εταιρείες που λένε ότι δεν θα δεν θα χρειάζονται μεγάλες, ε, μεγάλα εξαρτήματα ας πούμε, ε, μηχανών για να τυπώσουν αυτά που χρειάζονται. Επίσης, ε, υπάρχουν αθλητικά παπούτσια για το τρέξιμο, τα οποία κοσμήματα, διάφορα άλλα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν ε, την τεχνολογία της εκτύπωσης, ε, αθλητικά παπούτσια κτλ. Επίσης, αυτόνομα οχήματα, ε, μεταφράσεις από μηχανές, εφαρμογές στην αμυντική βιομηχανία. Όλα αυτά αλλάζουν τα δεδομένα για το γραφείο μας. Υπάρχουν πολλές αιτήσει για τους εξεταστές τεχνική νοημοσ... τεχνητή νοημοσύνη είναι στρατηγική σημασία και θα οδηγήσει σε τεχνολογικέ ε, εξελίξει και αλλαγέ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και οικονομικά και ηθικά θέματα. Είναι ένα τομέα που πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα, να καταλάβουμε τις, ε, το δυναμικό του, αλλά και να είμαστε προσεκτικοί, ειδικά σε ό,τι αφορά τα θέματα προστασία των δεδομένων που έχουν προκύψει, παραδείγματο χάρη το Facebook πρόσφατα. Ε, το γραφείο χρησιμοποιεί τα μεγα τα big data, τα μεγάλα δεδομένα, ε, για να σεβαστεί τους κανόνες ε, προστασίας των ε, δικαιωμάτων ιδιωτικότητας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες με σεβασμό των δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μείνει πίσω και να την ξεπεράσουν καλύτεροι ανταγωνιστές. Οι Αμερικάνοι, οι Ιαπωνέζοι κτλ. Ε, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και οι εφευρέσεις από την Κίνα και την Νότια Κορέα, ας πούμε. Ε, επίσης, πέρυσι οι αιτήσει για το εμπορικό σήμα από την Κίνα ε, διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2015 και η Κίνα είναι η τρίτη ε, μεγαλύτερη χώρα χρηματοδότηση μετά την Γερμανία και τις ΗΠΑ. Ε, το πρώτο τρίμηνο φέτος ε, οι αιτήσει ε, από την Κίνα ήταν αρκετές ε, και κάποιους μήνε μάλιστα ήταν και περισσότερε από τους Αμερικανούς. Ε, έχουμε μια μεταφορά ε, προς τα δεδομένα και, στις, και στα downloads. Και αυτό είναι τεράστια πρόκληση. Αυτά τα θέματα ε, τονίζονται σε διάφορες μελέτες του γραφείου ε, μέσω της δραστηριότητα του παρατηρητηρίου ε, και ο ΣΑ είπε ότι οι παραβιάσεις δικαιωμάτων δημοτικής ιδιοκτησίας στο διεθνές εμπόριο θα μπορούσαν να φτάσουν το 5% των ε, εισαγωγών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 88 δισεκατομμύρια το χρόνο. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη. Σε μια εποχή όπου το γραφείο θα πρέπει να, να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ζήτηση για νέα δικαιώματα ε, με πολλές αιτήσει που έρχονται από το εξωτερικό. Μία λύση είναι να καταλάβουμε καλύτερα τις τεχνολογίες που εμπλέκονται και να τις χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά για να ε, καταλάβουμε αυτόν τον περίπλοκο κόσμο. Θερυπίν. υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στα κρυπτονομίσματα και στο bitcoin. Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες πιθανές εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain ε, μερικές από αυτέ θα μπορούσαν να βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε τι παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία. Για να διευκολύνουμε την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, το γραφείο ε, στρέφεται στην Επιτροπή Προγραμματισμού και κωδικοποίηση ε, που γνωρίζουν πολύ καλά τι προκλήσει και το δυναμικό του blockchain. Το περασμένο μήνα το γραφείο ξεκίνησε μία, έναν διαγωνισμό τετραήμερο για να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το blockchain και να ενοποιήσουμε τις, τα συστήματα αξιών ε, μιλάμε, θα γίνει μάλλον τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες ε, και το βραβείο θα είναι 100.000. Ε, επίσης, ε, θα υπάρξει και ένα πρωτότυπο από, αυτή την, ε, το διαγωνισμό που ελπίζουμε να γίνει πραγματικό προϊόν. Ε, γνωρίζουμε πολύ περισσότερα τώρα για αυτά τα θέματα και το γραφείο ε, συνεργάζεται μαζί με άλλου ε, ε, φορεί μέσω του παρατηρητήου, ούτω ώστε στο μέλλον να δοθεί προτεραιότητα σε δραστηριότητε που υποστηρίζουν ε, επιτυχημένε προσπάθειε και που δίνουν τελικά απτά αποτελέσματα. θα πρέπει να δημιουργήσουμε εργαλεία, δίκτυα, να διευκολύνουμε τη συνεργασία με διάφορου φορεί, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε ένα πιο ενοποιημένο σύστημα. Πρέπει να επιμεριστούμε τα ε, δεδομένα και να βοηθήσουμε αυτούς που δημιουργούν τα δεδομένα. Θα ξέρετε ότι τα διάφορα εργαλεία εφαρμογή που έχει δημιουργήσει το εργαλείο, ε, βάσει δεδομένων εφαρμογή, ε, εργαλεία ε, κατά των απομιμήσεων και διάφορε βάσει δεδομένων για την ε, αναφορά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων σε τρίτε χώρε έχουν όλα ενοποιηθεί σε μία ενιαία πλατφόρμα το γραφείο μέσω του παρατηρητηρίου θα συνεχίσει να εργάζεται άμεσα μαζί με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς και γενικές διευθύνσεις ε, για να ε, διευκολύνει ε, την προσπάθεια καταπολέμησης του εγκλήματος μέσω της υπηρεσίας IPC. Το IPC 3 έχει λειτουργήσει για να κλείσει παράνομα online, παράνομες online αγορές και σχετική χρηματοδότηση. Κατέστρεψε επίση και διάφορε άλλε παράνομε προσπάθειε. Έχει κλείσει πολλέ ιστοσελίδε που προσφέρουν παραπημένα προϊόντα πολυτελεία, αθλητική ένδυση, ηλεκτρονικά, φάρμακα κλπ. Άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι είναι ισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των διαφερόμενων ε, με την πληροφορική ότι θα πρέπει να βοηθήσει το pc όταν έχουμε να κάνουμε με πειρατεία και απαραπημένα προϊόντα. Είναι ζωτική σημασία σε αυτή η προσέγγιση αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα εξαιτία της τεχνολογίας. Αλλά να ξέρετε ότι με κοινή προσπάθεια της υπηρεσίας μας και της Europol, Γενικών Διευθυντών και διαφόρων υπηρεσιών, Όλαφ, Γενικής Διεύθυνσης Ταξούτ και τα λοιπά, έχουμε αποτελέσματα. Και για πρώτη φορά υπάρχει μια τέτοια συνάντηση υψηλού επίπεδου για να συζητήσει ακριβώς αυτήν την ενισχυμένη συνεργασία για την καταπολέμηση της παραπής προϊόντων οι συμμετέχοντες είπαν πόσο μεγάλη σημασία έχει η ανταλλαγή απόψεων και η κοινή ανάλυση αλλά και η ενισχυμένη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εθνικές αρχές. Συγκεκριμένα μέτρα χρειάζονται για να καταπολεμηθούν οι παραβιάσεις πιο αποτελεσματικά. Συζητήθηκε αυτό το θέμα και οι συμμετέχοντες είπαν ότι θα ήθελαν τέτοιες συναντήσεις σε τακτική βάση και να τεθεί ένα πλαίσιο για να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει πρόοδο. Έγιναν οι μελέτες, ξέρουμε τα γεγονότα. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δράση. Τέτοιες συναντήσεις μπορούν να βοηθήσουν σε μια εξέλιξη όπου να καταλήξει σε μια συνολική στρατηγική. Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, το Γραφείο δημοτικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εξελιχθεί πολύ από το 2011 που σας συμβουλεύτηκε. Έχουμε καθορίσει τις προτεραιότητές μας και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις. Κοιτώντας πίσω, βλέπουμε ότι υπήρξαν κάποιες συγκεκριμένες τάσεις που βοήθησαν στην ε, πρόοδο και από τις οποίες θα εμπνευστούμε για το μέλλον. Πρώτο, πρέπει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας να γίνονται σεβαστά και να βοηθήσουμε γι' αυτό και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, πρέπει να γίνει κατανοητό το θέμα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Είναι δύσκολο βέβαια να προβλέψουμε τη στρατηγική μας επειδή αλλάζουν πολύ τα δεδομένα. Οι εξελίξεις τρέχουν με μεγάλους ρυθμούς. Πάντως, όλοι θέλουμε να προχωρήσουμε με μια αποκοινού κατανόηση της κατάστασης και να μπορούμε, αν μη τι άλλο, να ανταποκριθούμε στο βηματισμό των εξελίξεων. Η δικιά σας Επιτροπή μπορεί να μας βοηθήσει αποτελεσματικά να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές προκλήσεις. Όπως έχω πει πολλές φορές μέχρι τώρα, το σύστημά μας είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να προσφέρει ωφέλη στην οικονομία και στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που συνεχίζετε να δείχνετε ενδιαφέρον για το έργο μας και να παρακολουθείτε τις εξελίξεις ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί και τον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ. So, uh, thank you, Mr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καμπίνος για την τόσο πλούσια παρουσίασή σας. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο για ερωτήσεις. Ο κύριος Καβαντά πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω δημόσια να πω σε όσους βρίσκονται εδώ και σε όσους διαβάσουν τα πρακτικά πόσο χρήσιμο είναι το έργο του εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου Ιδιωτική Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πραγματικά προστατεύει την δημιουργία, τον πλούτο αυτό της δημιουργίας και των δημιουργών. Πολύ συχνά, λέω κάτι το 2014, που ετοίμασε μια ανεξάρτητη υπηρεσία, άρα την πιστεύουμε, που θύμισε τότε ότι ο δημιουργικός πλήτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάθε χρόνο πάνω από 531 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία ζουν πάνω από 7 εκατομμύρια άνθρωποι, ανεξάρτητα βέβαια από την καταστροφή που έχουμε από την παραποίηση προϊόντων. που τα παραβημένα προϊόντα μπαίνουν ε, από τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου είπανε πρόσφατα πόσα βαγόνια μπαίνουν σε μια χώρα ανατολικά της Επίρους μας και δυστυχώς οι χώρες μέλη δεν έχουν στη διάθεσή τους αρκετά εργαλεία για να το καταπολεμήσουν. Δεκάδες τρένα που έρχονται με προϊόντα από την Κίνα. Αυτό δίνει μια ιδέα για το τι προσπάθεια πρέπει να κάνουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τώρα. Τώρα που έχουμε την απόδειξη ότι το γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας λειτουργεί και έχουμε καλή πληροφόρηση. Θέλω να πω στους ε, εκπροσώπους του Κοινοβουλίου που στη δικιά σας συνέλευση εκπροσωπούν το σώμα. Δεν είμαι μόνος και ο κύριος Ιεύκα και η κυρία Λεγκρή που τώρα έχει πάει στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, αλλά και άλλοι. Θέλω να πω λοιπόν στους συνεδέρφους ότι περάσαμε από ένα στάδιο πολύ σημαντικού εξυγχρονισμού υπό την ηγεσία σας και με εξέπληξε το καλό αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες απομακρυσμένες από το κεντρικό πυρήνα και τώρα έχω την αίσθηση ότι βρίσκομαι μέσα σε ένα σώμα που λειτουργεί με πολύ σύγχρονο τρόπο και μπόρεσε η ομάδα σας να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στις εξελίξεις, κάτι που δεν ήταν εύκολο. Άρα μπορώ να φανταστώ τη δυσκολία επανοργάνωσης. Πάντως και το δικό σας γραφείο και το παρατηρητήριο πιστεύω ότι είναι όργανα ζωτικής σημασίας. Και θέλω να πω προσοχή να μην αντιταθούμε στο έργο τους, να μην μειώσουμε τον προϋπολογισμό, ιδίως σήμερα που ξέρουμε ότι διάφορες εμπορικές δυνάμεις ε, εκτός Ευρώπης προσπαθούν να μας επιτεθούν. Στον παγκόσμιο ανταγωνισμό είναι ζωτική σημασία. Το μόνο μέσο ανάλυσης που έχουμε στη διάθεσή μας για να παρατηρήσουμε τις τάσεις να λειτουργεί καλά. Και έτσι ο κύριος Καμπίνος, το λέω να το ξέρουν και οι συνάδελφοι, εξελέγει ε, αυτοκρατορικά θα έλεγα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν αυτοκράτορα, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πατέντας. Πράγμα που δείχνει ότι εκτιμήθηκε το έργο σας στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την ε, ανταλλαγή απόψεων και για την παρουσίαση από πλευρά του Πρόεδρου. Και θα ήθελα να πω ότι με έχει εντυπωσιάσει αυτό που μας παρουσιάσατε, η εργασία της υπηρεσίας σας. Καταλαβαίνω ότι θεωρείτε ότι παρέχετε ε, υπηρεσία και θεωρώ ότι είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικό αυτό. Είναι λειτουργήμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτά που μα είπατε για την διάρθρωση τη υπηρεσία σα και είναι πιστεύω εξαιρετικό το γεγονό ότι δεν έχετε μόνο υπόψη στη δική σα υπηρεσία, αλλά το ότι λέτε ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται και πέρα από ε, τα του οίκου μας και πώς θα συνεργαστούμε και με τις άλλες υπηρεσίες, με τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα και για τις κοινέ πλατφόρμες που θα πρέπει να βρεθούν. Αυτό λοιπόν που με εντυπωσιάζει είναι αυτά που μας είπατε για τις ε, τεχνολογίες blockchain. Νόμιζα ότι η υπηρεσία σας παρέχει τέτοιες δυνατότητες. και ότι δίνει τα κίνητρα ανάπτυξης και χρήση τη τεχνολογία blockchain. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακά αυτά που μα είπατε. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση να σα πω. Μίλησατε για την ανταγωνισμό από την Κίνα ιδιαίτερα. Και αναρωτιέμαι, βάσει των παρτρήσεών σα, οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι είναι καλύτεροι επειδή είναι πιο καινοτόμοι. Ή η διαφορά είναι στην εμπορική αξιοποίηση στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση των καινοτομιών. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε στον τομέα της καινοτομίας, της εκπαίδευσης ή δεν, ή αξιοποιούμε εμπορικά αυτά που ήδη έχουμε. Και στις παρατηρήσεις θα ήθελα να πω αυτό που είπε και ο συνάδελφος Καβαντά. Η δημιουργική βιομηχανία της Ευρώπης ε, και το περιεχόμενο που διαθέτουμε είναι το σημαντικό και δεν θα σταματήσω να λέω και εγώ αυτό που λέει και ο κ. Καβατά ότι δεν μπορούμε να διατεθούμε όλα δωρεάν στο διαδίκτυο θα πρέπει αυτή η παραγωγή, η δημιουργή να έχουν μια ανταμοιβή και άρα όλα όσα έχουμε φτιάξει στον τομείο του IPR έχουν να κάνουν και με την περιφερειακή ανάπτυξη της οικονομίας μας τελικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Είμαι από αυτούς που δεν κατάφερε να βρεθεί επιτόπου αλλά να ξέρετε ότι κάθε φορά που συζητάμε για το τι είδαν αυτοί που πήγαν στο Αλικάντε, τι συζητήθηκε, να ξέρετε ότι όλοι είναι ενθουσιώδεις εδώ στην Επιτροπή μας. Δηλαδή αυτό έχω εισπράξει εγώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Για το blockchain, μια σύντομη ερώτηση. Αναφέρθηκε και η Αγγέλικα Νίμπλερ στις τεχνολογίες αυτές. Μπορείτε να μπείτε περισσότερο σε βάθος Κάτι είπατε για τον Ιούνιο. Τι κάνετε για να αντιμετωπίσετε τις παραβιάσεις διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο κύριος Βιευσκά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως και οι προηγούμενοι, ιδιαίτερα ο κύριος Καβαντά. Έτσι και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τις προσπάθειες που έχετε κάνει μέχρι τώρα ως διευθυντής στο Αλικάντε. Αγαπητά Αντώνιο, εγώ έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια τις προσπάθειές σας από κοντά. Όταν, όταν ξεκινήσατε επικεφαλής εκεί στο Αλικάντε, που πιστεύω ότι είναι ένας από τους οργανισμούς που είναι καλύτερα οργανωμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ένα σωρό παραδείγματα καλής συνεργασίας που έχετε σχεδιάσει σε διεθνές επίπεδο. Είναι πραγματικά ένας από τους λίγους οργανισμούς που δεν μας κοστίζει. δεν το παίρνουμε είδηση οικονομικά. Κι όμως το έργο του προσφέρει πολλά ωφέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι λοιπόν που ο κύριος Καμπίνος τώρα πηγαίνει στο Μόναχο στη, στον οργανισμό πατέντας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ στους καιρούς που έρχονται. Όποιος και να σας αντικαταστήσει πάντως, θα είναι πολύ τυχερός μετά από τις προσπάθειες που έχετε κάνει εσείς στο Αλικάντερ. Η μόνη ανησυχία που έχουμε όλοι είναι ότι μπροστά μας υπάρχουν νέες προκλήσεις, γιατί αλλάζει η τεχνολογία περίπου σε καθημερινή βάση και εξελίσσεται. Οπότε η αντικατάστασή σας έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε τι θα γίνει με τη συνεργασία με τα όργανα εκείνα τα οποία ερευνούν τις παραβιάσεις που γίνονται σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι χώρες μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από τις έρευνες αυτές. Οπότε η ερώτησή μου είναι γιατί χάνουμε τη μάχη με τους Αμερικανούς και με τους ε, ασιατικούς Τίγρεις. Γιατί χάνουμε ιδέες και ταλέντα. Μήπως δεν προστατεύουμε αρκετά τα συμφέροντά μας και τα προϊόντα, τα δικά μας. μου φτάνουν κάποια νέα, ακόμα και από τη δικιά μου τη χώρα, την Πολωνία, προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάντως και για τη σκέψη σου. όσον αφορά τα βραβεία βρεσιτεχνίας των διαφόρων χωρών. Ελπίζω ότι οι δικές σου καλές πρακτικές θα βοηθήσουν, θα αποφέρουν καρπούς και στο μέλλον και ελπίζω ότι θα συνεχίσετε τις προσπάθειες και στο Μόναχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια πρώτα απ' όλα και για τις ερωτήσεις σας. Θέλω να απαντήσω, είναι βέβαια δύσκολο. Θα λέγα το εξής. Αν Κοιτάξτε, το επίπεδο επιστημονικών ε, άρθρων και τα λοιπά που δημοσιεύονται από ερευνητέ, καθηγητέ πανεπιστημίων και τα λοιπά, δεν βρισκόμαστε πίσω από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ούτε από του Κινέζου, καθ' Και έτσι έρχομαι στο συμπέρασμα ότι δεν είναι θέμα παραγωγής γνώσης, δεν υστερούμε σε αυτό από τους Αμερικανούς, είναι πώς τη γνώση αυτή θα τη μετατρέψουμε σε προϊόντα και σε καινοτομία για να έχουμε κέρδος στην αγορά και απασχόληση. Οι Αμερικανοί έχουν δύο πλεονεκτήματα σε σύγκριση με μας. Πρώτα απ' όλα είναι μία μόνο χώρα. Ενώ εμείς είμαστε ακόμα 28. Παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, εξακολουθούμε να είμαστε 28 διαφορετικές χώρες με διαφορετικά επίπεδα οριμότητας. Οι βόρειες χώρες, για παράδειγμα, ξέρουν και μεταφέρουν πολύ καλά τη γνώση και την κάνουν προϊόντα. Η Γερμανία κάνει πολύ καλά πράγματα. 19ο, 20ο αιώνα ήταν η καλύτερη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Οπότε αυτό που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε στο μέλλον περισσότερο είναι να κοιτάξουμε πώς λειτουργεί ολόκληρο αυτό το οικοσύστημα. Δηλαδή πώς ιδέες φτάνουν στην αγορά ε, πώς θα εντοπίσουμε τα καλύτερα παραδείγματα, ε, να εντοπίσουμε και τα κενά και να τα καλύψουμε. Χάσαμε την αρχή της επικουρικότητας που ήταν και η ομορφιά της Ευρώπης. Αυτό θα ήταν ένα στοιχείο. Λοιπόν, οι Αμερικανοί όντως είναι πάρα πολύ καλοί στο να μετατρέψουν τη γνώση, τις ιδέες σε προϊόντα, σε αγορά. Αυτό το κάνουν πολύ καλά. Και εμείς δεν πρέπει να μείνουμε στον αντοπισμό των προβλημάτων, αλλά να βρούμε και λύσεις. Οι Αμερικάνοι όντως φτιάξαν ένα οικοσύστημα πιο ευνοϊκό για αυτά. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για μία χώρα, όχι για 28 όπως είμαστε εμείς, αλλά δεν είναι καλύτερη στη γνώση, είναι καλύτερη στο να μετατρέπουν τη γνώση σε αγορά. Ε, περίπτωση μπλακετών. Η βασική ιδέα είναι... Έχουμε τέσσερις προγραμματιστές που έχουμε τοπίσει, που τέσσερις μέρες θα δουλέψουν για να ε, φτιάξουν ε, κώδικες. Η τεχνολογία blockchain αυτό το οποίο προσφέρει είναι ότι από τη στιγμή της δημιουργίας του προϊόντος μέχρι την διανομή του, η εξέλιξη του προϊόντος αυτού ελέγχεται πλήρως. Συνεπώς ξέρεις. Από τη στιγμή που παράγεται το προϊόν, το παρακολουθείς μέχρι τη στιγμή που διανέμεται στην αγορά. Να δούμε. Αυτά στη θεωρία, να δούμε στην πράξη τι θα γίνει. Τώρα, το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι το πώς μοιραζόμαστε τα δεδομένα μεταξύ μας. Ας πούμε η πορτογαλέζικη αστυνομία, που ξέρω, όταν ε, βρουν, εντοπίσουν ένα προϊόν, το ταξινομούν διαφορετικά. Έτσι κι δεν μπορείς να ανοίξεις όλα τα κοντέινερ στο Ρότερνταμ, ούτε είσαι σίγουρος ότι θα πετύχεις το σωστό κοντέινερ. Οπότε το θέμα είναι πώς θα μοιραζόμαστε τις πληροφορίες μεταξύ μας και πώς θα τις χρησιμοποιούμε. Αν υπάρχει μία τάση να είμαστε σε θέση να την παρακολουθήσουμε. Δεν θέλουμε να εμποδίσουμε το εμπόριο. Γι' αυτό η ανταλλαγή πληροφοριών είναι ζωτική σημασία. Και είναι πιο εύκολο όσο περνάει ο καιρό. Και για μας βέβαια, αλλά και για τους απαταιώνες, έτσι. Είναι το παιχνίδι της γάτας που κυνηγά το ποντίκι. Νομίζω ότι απάντησα σε ερωτήσεις σας. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Καμπίνος, θα ήθελα να σας κάνω και δύο επιπλέον ερωτήσεις. Καταρχάς, Μία πολύ γενική ερώτηση. Αναφερθήκατε στην ε, τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι ξέρουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε θέση να συγγράψει άρθρα, να συνθέσει μουσική και ούτω καθεξής. Σύμφωνα με τη συζήτηση που κάνατε, φαντάζομαι, αποτελεί αυτό πρόκληση για την ορισμό των ίδιο του έργου του διανοητικού με προστασία διανοητικών δικαιωμάτων και αν ναι, πού οδεύει αυτή η συζήτηση στον IPO. Δεύτερη ερώτηση. Ο όγκος εφαρμογών και GI μη γεωργικής φύσης μας έχει αποδείξει ότι χρειάζεται τέτοιου είδους προστασίας. Κοιτάξτε, είναι όλο και πιο δύσκολο να απαντήσω στα ερωτήματά σα. Να ξεκινήσω από την δεύτερη ερώτηση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει μη γεωργική προστασία GI. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μελέτη αντικτύπου για το κατά πόσο χρειάζονται. Γιατί όπω σα είπα, το IP είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο δημόσιο ιδιωτικό κλάδο ή και όχι. Δεν θα καθορίσουμε εμεί κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Αυτό θα το αποφασίσει από μόνο του ο ιδιωτικό κλάδο. Αν δεν υπάρχει όμω το εργαλείο εξορισμού, δεν θα χρησιμοποιηθεί. Μη γεωργικά λοιπόν GI υπάρχουν εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, για παράδειγμα, που περιλαμβάνει πολλέ ε, εφαρμογέ και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μην περιμένουμε λοιπόν άλλο. Και κοιτώντα του ε, φίλου μου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πω το εξή. Όταν κάναμε τι ε, συμφωνίε ε, FTA, υποβάλαμε γεωργικά GIs. Για τις γεωγραφικές ενδέξεις, λοιπόν, Υπάρχει λοιπόν μια switch σε προστασία. Και μου είπανε, Αντώνιο, υπάρχει ε, κάπου μια αναφορά ενό trademark που περιλαμβάνει ε, μια γεωγραφική ένδειξη. Μου φαίνεται, μα δεν είναι τρόπος να δουλέψουμε αυτός για να χάνουμε χρόνο σε μελέτες αντικτύπου που έχουν γίνει ο κανόνας για να καθορίσουμε κατά πόσο υπάρχει ο ελέφαντας στο, στην αίθουσα, νομίζω ότι είναι ε, ε, απώλεια μη χάνουμε χρόνο. Όταν υπάρχει ο ελέφαντα στο δωμάτιο, απλά να γνωρίσουμε ότι υπάρχει. Για την πρώτη ερώτηση τώρα. Δεν φταίει πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε πολλές περιπτώσεις φταίμε και εμείς και φταίνε και όλοι. Για την άλλη ερώτηση. Το copyright. Ο κανονισμός θα καταλήξει μετά από επίσημη απόφαση. Ναι, δεν μας απασχολεί πάρα πολύ, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται με τέτοιους ρυθμούς που το iPay, το οποίο έχει δημιουργηθεί στο τέλος του 19ου αιώνα και στον 20ο αιώνα, πλέον διακυβεύεται. Θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Αλλά Υπάρχουν ε, πολλά ερωτήματα που δεν έχουν ακόμα απαντηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε τα trademarks, τα εμπορικά σήματα. Έχουμε και τα κινητικά σήματα. Δεν έχει τροποποιηθεί όμως ο κανονισμός για το σχεδιασμό. Ο σας είπα και δεν ήσασταν εδώ πέρα. Μπορεί να προστατεύσουμε λοιπόν με τον κανονισμό αυτό στην Κορέα, αλλά όχι στην ε, Ευρώπη έργο. Χάνουμε λοιπόν δυναμικό, πιστεύω ότι ναι. Ξεκάθαρα. Και κοιτώντας λοιπόν τι διακυβεύεται εδώ, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της βιομηχανίας, το θέμα των αρκτικών. Αυτό μπλοκάρει τις αλλαγές στον ε, κανονισμό για το σχεδιασμό. Γιατί όλοι φοβόμαστε για τα ανταλλακτικά. Κάποια κρατημέλη πιστεύουν ότι πρέπει να πάμε προς τη μία και κάποια άλλη προς την άλλη. Αλλά χάνουμε. Λόγω της συζήτησης αυτής, η οποία θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει ξεχωρίστα, ε, χάνουμε την ευκαιρία να εξυγχρονίσουμε τον κανονισμό για το σχεδιασμό. Είναι από το 2003 πρέπει επιτέλου να ενημερωθεί. 18 έχουμε φτάσει. κοινοτική, λοιπόν, κοινοτικό σχεδιασμό, όχι ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Μην με ρωτήσετε μόνο άλλε ερωτήσει. Εν συντομία. Την προηγούμενη εβδομάδα συνέβη κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να διδαχθούμε από αυτό. Είπατε πριν από λίγο πόσο σημαντική είναι η προστασία των πληροφοριών, των δεδομένων, αυτή αποτελεί τη βάση του διαρκή εμπλουτισμού και των ε, επιχειρήσεων που δεν μπορούν να αφήνουν να ξεφεύγουν αυτά τα στοιχεία. Αυτό λοιπόν που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα είναι το εξή. Η, η ε, που προστατεύει τα προσωπικά της δεδομένα, μάλλον η ΕΠΑ, σε ό,τι αφορά την Αμερικανική Γερουσία και το Κογκρέσο, τι ακούσαμε, μεγάλο μάθημα. Ο δρόμος που και αυτά που είπαν οι Αμερικανοί ηθήνοντες που είπαν ότι τελικά η Ευρώπη προστατεύει καλύτερα τα δεδομένα της. Το λέω αυτό όχι για να κατηγορήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά για να την ενθαρρύνω και ποιοτικά και ποσοτικά να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπως οι χώρες του Περσικού κόλπου μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Έχουμε κάποια στοιχεία, αλλά δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Και αυτοί υποφέρουν στην Ευρώπη είναι αυτή το περιθώριο ε, εμπλουτισμού και κέρδους ε, που έχουμε θα πρέπει να το προστατεύσουμε. Αν ε, ακόμα και οι Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστοί για τις κολακίες τους προς τους Ευρωπαίους, αναφέρουν ότι τα πληρώνουν καλύτερα, θα πρέπει κάτι να σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Έχω 14 λεπτά για να επαναλάβω τους επένους. Προς το πρόσωπό σας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ από πλευρά της Επιτροπής μας για όλο το χρόνο που μας αφιερώσατε για ανταλλαγή απόψεων. όλα αυτά τα χρόνια. Ε, είμαστε πολύ ευγνώμονε γιατί πάντα ήταν πολύ επικοδομητική η ανταλλαγή απόψεων και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η παράδοση όσο θα είσαστε στη θέση σας ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσία για τις Ευρεσιτεχνίε. Γιατί και αυτό, αυτή η υπηρεσία συγκαταλέγεται στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας δεν θα σας χάσουμε λοιπόν, δεν θα χαθούμε και προσβλέπουμε να ακούσουμε από εσά και υπό τη νέα σας ιδιότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, κοιτάξτε, για να μην έχω προβλήματα όταν φτάσω στο Μόναχο, όπως ξέρετε το EPO είναι Ευρωπαϊκή Δημόσια Υπηρεσία, αλλά δεν είναι στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχετε νομική αρμοδιότητα για μας, αλλά με μεγάλη χαρά θα έρθουμε στην Επιτροπή σας. Μάλιστα, είσαστε πολύ ακριβεί. και σωστός. Αλλά η ανταλλαγή απόφαση, οι ανταλλαγέ ε, απόψεων με την Επιτροπή μας ε, είναι μία από τι καλέ παραδόσει που έχουμε, εν περιπτώσει.